τη μέση διάταξη. Ευχαριστώ. επόμενο σημείο. Ανακοινώσεις της Προέδρου. Όπως γνωρίζετε, οι πιο πολλές ε, ε, ανακοινώσεις θα αφορούν την Αφρικανική Εβδομάδα στο Αμπιτζάν. Την επόμενη εβδομάδα έχουμε την διάσκεψη κορυφή Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και Αφρικής πολύ σημαντική συνάντηση όπου θα επαναξιολογήσουμε τις σχέσεις της Ένωσης με την Αφρική και σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος Ταγιάννη αυτή την εβδομάδα ε, θέσπισε την Αφρικανική Εβδομάδα εδώ στο Κοινοβούλιο. Έχουμε πολλές δραστηριότητες και τις δικές μας, ε, τη δική μας συνεδρίαση σήμερα και άλλες δραστηριότητες. Να υπενθυμίσω ιδίω στου συνεργάτε ε, να ενημερώσετε του βουλευτέ σα, γιατί αύριο το πρωί έχουμε μια κοινή συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Θα συζητήσουμε του στόχου τη βιώσιμη ανάπτυξη. Από 24 χώρε έχουμε ομολόγου μα από τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και θα συζητήσουμε μαζί του την υλοποίηση των στόχων τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θα έχουμε από τον Ιγυριανό Κοινοβούλιο προσκεκλημένου λοιπόν, και από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο Επίση, έχουμε κάποιου συναδέλφου. Πολύ σημαντική συνάντηση αύριο. Ελπίζω να είναι μεγάλη προσέλευση και παρακαλώ τους συνεργάτε των πολιτικών ομάδων να ενημερώσουν τους βουλευτέ. Γιατί σημαντική αυτή αυριανή συνεδρίαση. Επίσης, αύριο στις 2.30 ε, στην Επιτροπή περιβάλλοντο, έχουμε αντιλαγή απόψεων, παρότι συμπίπτει εν μέρη, με τον δόκτορα Μοέτη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και το μεσημέρι που δεν συνεδριάζουμε, άρα μπορούν να πάνε συνάδελφοι, από τις 7 παρατέταρτο έως τις 8 παρατέταρτο, μια ειδική συνεδρίαση της Ομάδας Υποστήριξης Δημοκρατίας που επιβλέπει στο Κοινοβούλιο, τις αποστολές εκλογών, παρατήρησης εκλογών και το έργο μας που αφορά την δημοκρατία με χώρες εταίρους και το θέμα θα είναι οι εκλογές στην Αφρική, εστιάζοντας ιδίω στις εκλογές στην Κένια. Αλλά θα δούμε και τα ευρύτερα ζητήματα που άπτονται της δημοκρατίας στην Αφρική. Με ενδιαφέρουσες εξελίξεις, όπως ξέρετε, τις τελευταίες μέρες στη Ζιμπάμπουε. Πολλά έχουμε να πούμε λοιπόν. Όλα αυτά αύριο το απόγευμα. 7 παρατέταρτο με 8 παρατέταρτο το απόγευμα στην αίθουσα ΑΣΠΑ 1Ε2. Γράψτε το και αυτό παρακαλώ για να ενημερώσετε τους βουλευτές. Πολλά γίνονται, αλλά να τους υπενθυμίσουμε. Τουλάχιστον σίγουρα να έρθουν αύριο το πρωί στην συνάντηση μας με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Και βέβαια έχουμε και μία διάσκεψη ψηλού επίπεδου που λέγεται Ανανεωμένη εταιρική σχέση με την Αφρική. Αρχίζει την Τετάρτη στις 2 το μεσημέρι στο ημικύκλιο. Και υπάρχουν ε, και τρεις ε, γύροι τραπεζών, θα εκπροσωπηθούν ε, σημαντικοί φορείς από τις αφρικανικές χώρες και ο πρόεδρος Ταγιάννη που είναι ο χορηγός. Θα είναι εκεί. Δεν έχετε να πείτε κάτι. Πάμε στο σημείο 3 που είναι η των πρακτικών, συγκεκριμένα τη συνεδρία τη 31η Αυγούστου. Είναι στο φάκελό σα τα πρακτικά. Αν έχετε παρατηρήσει, στείλτε τα στην ΑΝ, στην γραμματεία πριν το τέλο τη συνεδρίαση. Και αν δεν έχουν παρατηρήσει, θεωρούμε ότι θα έχουν, θα θα έχουν εγκριθεί. Πάμε στο σημείο 4, ανακοινώσει ε, τη Επιτροπή. Κάποια ανακοίνωση νομίζω υπάρχει. Ποιο θα την κάνει. Ευχαριστώ πολύ. Σύντομη ενημέρωση κατόπιν μια προηγούμενης ανακοίνωση. Aid for Trade Communication. Η εν λόγω ανακοίνωση έχει ένα πολύ μακρύ τίτλο βέβαια. Έχει κοινοποιηθεί επισήμω ε, στου ε, ενδιαφερομένους. You put it on your radar. Απλά σας το λέω να έχετε υπόψη σας. Και μπορούμε να έρθουμε να συζητήσουμε την ανακοίνωση αυτή σε μια προσεχή συνάντησή σας. Ναι, πράγματι το έχουμε και στις συνεδρία των συντονιστών. Να δούμε την νέα ανακοίνωση του Aid for Trade, πώς θα την χειριστούμε. Σημαντικά ζητήματα για το επόμενο εξάμεινο. Θα τα δούμε. Περνάμε στο σημείο 5. Πρώτο σημείο για την Αφρικανική Εβδομάδα. Θα έχουμε και τη UNICEF εδώ, χαίρομαι πολύ, που έχουν εκπονήσει μια έκθεση για τη γενιά 2030 Αφρική. Προτεραιότητα σε επενδύσει στα παιδιά για την αντιμετώπιση του δημογραφικού ελλείμματος. Σήμερα είναι η Οικομενική Μέρα του Παιδιού. είχε εγκριθεί την ίδια ημέρα η διακήρυξη των ΗΕ για τα δικαιώματα των παιδιών. Και για τους Ροχίνγκα το Σαββατοκύριακο, ε, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις ε, βλέπουμε ότι τα δικαιώματα των παιδιών δεν γίνονται σεβαστά. Προσβλέπω στη σημερινή συνάντηση. Δεν ξέρω αν έχετε αντίτυπα αυτής της έκθεσης. Τα έχετε στείλει. Ποιο είναι από τα δύο αυτό. Generation 2030 Αφρικα. Έχετε αντίτυπα. Έχεις, Σάρλ, όχι. Λοιπόν, να διαθέσουν παρακαλώ, να, δια... να μοιράσετε παρακαλώ αντίτυπα από το έγγραφο της UNICEF στους βουλευτές. Μια σημαντική έκθεση αυτή. Έχουμε εδώ την Μπάρμπαρα Μπεντέ. Α, δεν έρχεται. Την Σάντι Μπλάνσετ. Ναι. Η κυρία Μπλάνσετ θα μας παρουσιάσει τη μελέτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα πάρετε εσείς καταρχάς το λόγο. Um, thank you very much, Madam Chair. Uh, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Είναι μεγάλη μου χαρά που βρίσκομαι εδώ σήμερα για να σας παρουσιάσω αυτή την έκθεση για τη γενιά του 2030 με αισθήσει στην Αφρική. Στην Αφρική και στα παιδιά και στους νέους ανθρώπους της Αφρικής. Όπως είπατε κυρία Πρόεδρε, η μέρα αυτή είναι ιδιαίτερη. Είναι η Παγκόσμια Μέρα των Παιδιών και ε, σε ολόκληρο τον κόσμο θα υπάρξουν ε, διάφορες εκδηλώσεις για την πρόθεση και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Φυσικά όλη η εβδομάδα αυτή είναι αφιερωμένη στην Αφρική συντονίζονται όλα αυτά και χαίρομαι που είμαι εδώ για να σας μιλήσω για την Αφρική από απόψη ε, δημογραφική, γενεολογική και να σας μιλήσω ειδικότερα για τα Παιδιά, ξέρετε ότι η Σύνοδος Κορυφής ε, στην Αφρική θα εστιαστεί στους νέους. Ξέρετε, οι άνθρωποι δεν γεννιούνται στην ηλικία των 15, ούτε πέφτουν από τα δέντρα, πρέπει να γεννηθούν, να εμβολιαστούν, να μορφωθούν ε, και να προστατεύονται. Οπότε θέλουμε να εστιαστούμε στις ηλικίε ομάδες από 0 μέχρι 18. Μια επένδυση που πρέπει να απασχολήσει την Αφρική και τους εταίρους της. Έτσι θα διασφαλιστεί ότι η Αφρική θα αξιοποιήσει το δημογραφικό μέρεσμα. Το δημογραφικό μέρεσμα αφορά μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή στην εξέλιξη μιας χώρας. Είναι η στιγμή όπου ο ενεργός πληθυσμός, οι εργαζόμενοι ενήλικες, υπερβαίνουν σε αριθμό τον ενεργό πληθυσμό. Συνήθως ε, αναφερόμαστε εδώ σε παιδιά και σε ηλικιωμένους. Και επειδή ο ενεργός πληθυσμός ε, είναι μεγαλύτερο μεγέθους, τότε η χώρα, η Ήπειρος ε, που συζητάμε, μπορεί να σημειώσει γρήγορη εξέλιξη. Η εμπειρία των τελευταίων 200 ετών δείχνει ότι αυτό το δημογραφικό μέρισμα μπορεί να αποδειχθεί εποφελές μόνο εφόσον έχουν γίνει επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Δηλαδή μόνο εφόσον έχουμε επενδύσει σε παιδιά, στην παιδεία τους, στην υγεία και στην προστασία τους. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τους ε, βιώσιμους στόχους της για το 2030, με τους, με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης του 2030 που εφαρμόζονται παγκοσμίω. Ήδη σήμερα τα παιδιά που τελούν σχεδόν το ίμιση του πληθυσμού της Αφρικής ε, μέχρι το 2030 θα έχουν προσθεθεί σε αυτά 170 εκατομμύρια παιδιά στην Αφρική. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το 2030 ο παιδικός πληθυσμός στην Αφρική θα έχει φτάσει τα 750.000 παιδιά. Τεράστιος αριθμός που αποτελεί ταυτόχρονα μια τεράστια ευκαιρία αλλά και μια τεράστια πρόκληση. Όπως είπα, αυτό που είναι σημαντικό για την Αφρική είναι να καταφέρει να αξιοποιήσει αυτό το δημογραφικό μέρισμα. Είναι σημαντικό να ξεκινήσουν τώρα οι επενδύσεις για τα παιδιά και να συνεχιστούν μέσα στα 15 χρόνια. Τα 15 χρόνια που θα ακολουθήσουν αποτελούν ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρία, ε, όπου θα πρέπει να εστιαστούμε στην υγεία, στην παιδεία και στην προστασία, την προστασία από τη βία και την κοινωνική προστασία. Υπό αυτόν τον όρο, μετά στις δεκαετίες του 30, του 40 και του 50 η Αφρική θα μπορέσει να βιώσει ε, σταθερή ανάπτυξη, ευημερία, ειρήνη και εξέλιξη. Η κατάσταση στην Αφρική έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία 30 χρόνια. Έχουν σημειωθεί τεράστιες πρόοδοι και μερικές φορές το ξεχνάμε, διότι συχνά οι ειδήσει για την Αφρική είναι μόνο κακές. Αυτό που θέλουμε να επισημάνουμε λοιπόν και το κάνουμε και στην έκθεσή μας ε, είναι ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος για τα παιδιά στην Αφρική. Ωστόσο, εξακολουθούμε να βλέπουμε ελλείψεις. Τρεις ε, που θεωρούμε σημαντικότερες είναι πρώτη η παιδεία. Μόνο για να διατηρηθεί ο τρέχον αριθμός μαθητών στα σχολεία στην Αφρική. Θα πρέπει να προσθεθούν 1,3 εκατομμύρια δάσκαλοι μες στην επόμενη δεκαετία. Αυτό όμως και πάλι δεν είναι επαρκές, διότι ε, πολλά παιδιά δεν ε, ολοκληρώνουν το, το, δημοτικό. Τι πρέπει να γίνει λοιπόν η Αφρική πρέπει να επενδύσει σε 5,8 εκατομμύρια προς δασκάλους για να ε, πληρεί τα διεθνή πρότυπα. Τα διεθνή πρότυπα που αναφέρονται εδώ στην έκθεση είναι 23 μαθητές ανά ένα δάσκαλο. Αυτό σημαίνει κατά βάση ότι την επόμενη 15 ετία η Αφρική θα πρέπει να διπλασιάσει τον αριθμό των δασκάλων, των διδασκόντων, ώστε να είναι βέβαιο ότι θα επιτύχει τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και ειδικότερα την ε, καθολική ε, εκπαίδευση δημοτικού και πρέπει επίση να γίνει κάτι και για τη δευτερεύουσα εκπαίδευση. Ξέρετε ότι πολλά παιδιά στην Αφρική πάνε στα σχολεία και δεν μαθαίνουν αρκετά. Είπανε σχολεία, μαθαίνουν κάποια πράγματα, αλλά αυτά δεν του ωφελούν για την εργασία. Οπότε πρέπει και η ποιότητα να ενισχυθεί, να αναθεωρηθεί το πρόγραμμα σπουδών σε πολλέ χώρε, η εκπαίδευση των δασκάλων, να αυξηθεί ο αριθμό των σχολείων, η ποιότητα των εγκαταστάσεων, ε, πιο συγκεκριμένα ξεχωριστέ τουαλέτε για και για κορίτσια. Ξέρω ότι οι αριθμοί αυτοί είναι τεράστιοι. Αν δούμε το παράδειγμα μιας χώρας, ε, μια χώρα που δεν ακούμε συχνά για καλέ ειδήσει, ε, τον Νίγηρα. Το Νίγη, στον Νίγηρα τα τελευταία 15 ετία η ολοκλήρωση των σπουδών δημοτικού έχει φτάσει το, από το 16% στο 59%. Είναι τεράστια η αύξηση για μόνο διάστημα 15 ετών. Η αιτίες ε, ήταν οι διαρκείς επενδύσεις από πλευράς κυβέρνησης και εταίρων της. Ο προϋπολογισμός, ε, ο κρατικός που εκχωρείται στην εκπαίδευση έχει ανέβει από το 17% στο 22%. Ο μισός προϋπολογισμός της ε, εκπαίδευσης πηγαίνει στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ώστε να είναι βέβαιο ότι τουλάχιστον όλα τα παιδιά θα πάνε και θα μάθουν κάτι. Ο αριθμός των σχολείων έχει διπλασιαστεί και ο αριθμός των διδασκόντων έχει τριπλασιαστεί. Στην παιδεία επίσης πρέπει κανείς να εστιαστεί και στην παιδεία των κοριτσιών. Όχι μόνο γιατί τα κορίτσια μένουν πίσω δυστυχώς, γιατί ξέρουμε ότι ο αριθμός ε, εγγραφής ε, κοριτσιών στο σχολείο είναι μικρότερος από των αγοριών, αλλά και γιατί η επένδυση στην ε, εκπαίδευση των κοριτσιών αποφέρει πολλά ωφέλη. Έχουμε στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι νέες κοπέλες, τα κορίτσια χωρίς ε, παιδεία, ε, κάνουν ε, κατά μέσο όρο 6,7 παιδιά, ενώ οι γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει την πρωτεύουσα εκπαίδευση αποκτούν κατά μέσο όρο 5,8 παιδιά. Και οι γυναίκες που έχουν ολοκληρώσει τις δευτεροβάθμιες σπουδές έχουν ακόμη μικρότερο μέσο όρο. Οπότε όσο πιο μορφωμένε είναι οι γυναίκες, όχι μόνο είναι πιο παραγωγικές ως εργαζόμενοι, αλλά κάνουν και λιγότερα παιδιά. Αυτό σχετίζεται και με τους ε, γάμους ε, ανηλίκων, γιατί όταν τα κορίτσια πηγαίνουν στο σχολείο, παντρεύονται πολύ αργότερα. Στον τομέα της υγείας, και εκεί έχει σημειωθεί κάποια πρόοδο, αλλά απαιτούνται περισσότερε επενδύσει. Εμείς χρησιμοποιήσαμε εδώ τα benchmark του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην έκθεσή μας ε, που είναι ο αριθμός εργαζομένων στον τομέα της υγείας ανά χίλιους ανθρώπους και στην Αφρική αυτή τη στιγμή ο μέσος είναι 1,7 επαγγελματίες ανά χίλιους ανθρώπους, ενώ στη Δανία, για να καταλάβετε ε, συγκριτικά, είναι 20 εργαζόμενοι στον τομέα υγείας ανά χίλια άτομα. Αν θέλουμε το 1,7 να πάει στο 4,45 που είναι το κατόφλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα χρειαστούμε πολλούς περισσότερους εργαζομένους στον τομέα της υγείας στην Αφρική. Ο αριθμός σήμερα ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια και αν συνεχίσουμε με τις σημερινές τάσεις θα φτάσουμε τα 2,4 εκατομμύρια μέχρι το 2030. Ωστόσο η μελέτη μας δείχνει ότι για να φτάσουμε στο πρότυπο του, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας χρειαζόμαστε επιπλέον 4,2 εκατομμύρια εργαζομένους στον τομέα της υγείας. Είναι τεράστιος αριθμός και φυσικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι πρέπει να εκπαιδευτούν και μετά να προσληφθούν και να διατηρηθούν στο σύστημα. Αλλά το παράδειγμα της Ρουάντα δείχνει ότι είναι δυνατό να σημειωθεί σημαντική πρόοδο στον τομέα της υγείας ε, η βρεφική θνησιμότητα ήταν 151 στους χίλιους ε, στην Ουγκάντα και έχει πέσει στο 39 μέσα σε μία γενιά. Αυτό έγινε με την επέκταση των κοινοτικών υπηρεσιών υγείας ε, με εστίαση ε, στην αγροτική παροχή υγείας ενισχύοντας τις δυνατότητες των αγροτών και παρέχοντας τους κίνητρα καθώς επίσης και με την ανάπτυξη ε, προγραμμάτων υγείας ε, κοινοτικής φύσης. Οπότε οι φτωχοί άρχισαν να αποκτούν περισσότερες υπηρεσίες υγείας ε, σε σχέση με τους λιγότερο φτωχούς. Όλα αυτά σχετίζονται και με την προστασία. Υπάρχει το ζήτημα τη βία κατά των παιδιών στην Αφρική. Δεν είναι μόνο η Ήπειρο φυσικά, αλλά είναι μια Ήπειρο όπου το φαινόμενο είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Όπω επίση και οι ανισότητε μεταξύ φύλων. Και αυτά τα δύο πράγματα είναι αλληλένδετα. Όταν μιλάμε για προστασία από τη βία, μιλάμε στο σπίτι, στην κοινότητα και στη χώρα. Είναι τρία τα επίπεδα. Πολύ συχνά οι γυναίκες και τα κορίτσια είναι τα ε, θύματα ε, κάθε μορφής βίας. Ε, οι παιδικοί γάμοι ακόμα αφορούν το 55% των γυναικών και των κοριτσιών στην Αφρική. 35%, το 35% των γυναικών σήμερα έχουν παντρευτεί πριν από τα 18 τους. Αλλά χώρες όπως η Μπουρκίνα Φάσο και η Αιθιοπία δείχνουν ότι είναι δυνατόν μέσω συντονισμένων και συνεχών προσπαθειών να μειωθούν οι γάμοι ανηλίκων όπως και οι ε, ακροτηριασμοί των κοριτσιών. το 46% δεν λαμβάνει πιστοποιητικά γέννηση, ε, ε, το οποίο δημιουργεί πρόβλημα αργότερα σε αυτούς τους ανθρώπους όταν μεγαλώσουν, αποτελεί εμπόδιο για να πάνε στο σχολείο, να βρουν δουλειά, να ανοίξουν ένα τραπεζικό λογαριασμό ή να ψηφίσουν. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι το 74% των παιδιών λαμβάνουν ε, τρεις δόσεις εμβολίων. δωρεάν, συγγνώμη, δόσεις εμβολίων. Οπότε, η πρόκληση εδώ είναι αντί να εργάζεται κανεί μεμονωμένα μόνο στον τομέα του με τα παιδιά, ε, ε, θα ήταν να έχουμε όλου αυτού του επαγγελματίε να συνεργάζονται. Οπότε, ας πούμε, οι εργαζόμενοι υγεία να διασφαλίζουν ότι θα παρέχονται και επιστοποιητικά ε, γέννηση σε παιδιά. Το 49% των παιδιών ζουν σε εξαιρετική φτώχεια στην Αφρική, δηλαδή με κάτω από 2 δολάρια ημερησίω. 49% μιλάμε για το μισό παιδικό πληθυσμό της Αφρικής σε σύγκριση με το 38% των ενηλίκων. Δηλαδή όχι μόνο η Αφρική υποφέρει από ένα πρόβλημα φτώχειας, αλλά τα παιδιά στην Αφρική είναι πιο φτωχά από ότι οι ενήλικες. Ξέρουμε τα παιδιά που γεννιούνται σε ακραία φτώχεια και που δεν έχουν πρόσβαση σε υγεία, παιδεία και διατροφή δεν θα να μεγαλώσουν κανονικά. Τα, τα σώματά τους, τα μυαλά τους δεν ε, ε, ε, οι ψυχοί του δεν θα αναπτυχθούν όπω των άλλων ανθρώπων και δεν θα φτάσουν στα επίπεδα παραγωγικότητα και συμμετοχή στην κοινωνία όπω ε, άλλοι άνθρωποι. Το 25% των παιδιών στην Αφρική ζουν σε χώρε ε, ε, συγκρούσεων ή σε εύθραυστο περιβάλλον. Αυτό αντιστοιχεί σε 153 εκατομμύρια παιδιά που κάθε πρωί ξυπνούν με το φόβο βίας, πολέμου, οργανωμένης βίας στις κοινότητες στις χώρες τους. Και φυσικά η κλιματική αλλαγή επίσης επηρεάζει την Αφρική όπως όλοι γνωρίζουμε πολύ περισσότερο από άλλες υπήρου λόγω ε, της μη θωράκησης των κοινοτήτων και των χωρών. Ε, δηλαδή το, ξέρουμε ότι πάνω από το 50% των παιδιών ε, ζουν σε περιοχές ε, που πλήττονται από ξηρασίες ε, μέτριας κλίμακας ή έντονες. Όλα αυτά συντονίζονται μεταξύ τους. Ένα παιδί που πάει στο σχολείο αλλά δεν τρέφεται καλά δεν πρόκειται να μάθει τόσο πολλά πράγματα. Ένα παιδί που πάει στο σχολείο πολύ συχνά ε, προστατεύεται από τη βία, όπως είπα προηγουμένως. Ένα κορίτσι που πάει σχολείο θα παντρευτεί αργότερα. Ένα παιδί υγιές που δεν έχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό είναι πιο πιθανό να αρρωστήσει. Ένα παιδί που πρέπει να περπατήσει 10 χιλιόμετρα για να πάει να βρει νερό για την οικογένεια, ειδικότερα τα κορίτσια, δεν θα έχει το χρόνο να πάει στο σχολείο. Οπότε πρέπει να λύσουμε αυτά τα προβλήματα όλα μαζί, επειδή είναι αλληλένδετα. Τώρα από πλευρά UNICEF ήδη επενδύουμε τεράστια ποσά στην Αφρική στα προγράμματά μας. Πέρυσι σχεδόν ο μισός μας προϋπολογισμός, δηλαδή 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, επενδύθηκαν στην Αφρική με εστίαση στα παιδιά και στις οικογένειές τους. Αυτή οι πόροι, αυτά τα χρήματα της UNICEF προέρχονται κυρίως από κυβερνήσεις, αλλά και από τα θεσμικά οργανά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τους Ευρωπαίους πολίτες, ε, τους ίδιους τελικά αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα και από ιδιώτες. Πολλοί, όπως είπαμε, Ευρωπαίοι πολίτες που δίνουν, να κάνουν δωρεές στη UNICEF, οπότε θα ήθελα να δράξω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω ε, τις κυβερνήσεις και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τη γενοδερία τους ε, προς υποστήριξη των παιδιών αυτών. Όπως είπα προηγουμένως, οι προκλήσεις είναι τεράστιες, αλλά γνωρίζουμε από χώρες που τα καταφέρουν ότι είναι δυνατό Έχουμε δει καλά παραδείγματα και στην Αφρική και στην Ασία και στην Ασία κατάφεραν να αξιοποιήσουν αυτό το δημογραφικό μέρεσμα. Πρόκειται για μια συζήτηση που θεωρούμε είναι πολύ σημαντική σε επίπεδο ε, Συνόδου Αφρικανικής Ένωση και Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να αδράξω την ευκαιρία για να υπενθυμίσω στι κυβερνήσει ότι είναι καθήκον του σύμφωνα με τη συνθήκη για τα δικαιώματα του παιδιού όλες οι που, την οποία έχουν κυρώσει όλε οι αφρικανικές και ευρωπαϊκέ κυβέρνησεις. Είναι υποχρέωση των κυβερνήσεων να επενδύσουν στα παιδιά, στην υγεία, στην παιδεία, στην προστασία του παιδιού και στην κοινωνική προστασία. Και θα ήθελα να, με την ευκαιρία να κάνω έκκληση, να απευθύνω έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Ένωση να επενδύσει το 20% της ανθρωπιστικής βοήθειας ε, στους τομείς αυτούς. Ε, αυτό αναφέρεται και στην έκθεση του κυρίου Πόγκα για τις σχέσεις Αφρικανικής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη UNICEF ε, πιστεύουμε ότι υπάρχει ηθική και νομική υποχρέωση να υποστηρίξουμε τις επενδύσεις στα παιδιά. Ακούμε συνέχεια γύρω μας ότι συμφέρει τόσο την Ευρώπη όσο και την Αφρική να επενδύσουν στα παιδιά και στους νέους ανθρώπους στην Ήπειρο αυτή. Πιστεύω ότι όλοι μαζί έχουμε αυτή την ευκαιρία να κάνουμε τη διαφορά, να επιταχύνουμε την πρόοδο για τα παιδιά της Αφρικής, αλλά και για ολόκληρη την Ήπειρο και σε τελική ανάλυση ε, για όλο τον κόσμο, διότι οι στόχοι βεσμής ανάπτυξης δεν πρόκειται να επιτευχθούν χωρίς την Αφρική. Ευχαριστώ πολύ. Έπρεπε να πω, ότι, ε, έπρεπε να πω εξ αρχής ότι η Σάντι είναι διευθύντρια του γραφείου της UNICEF και είναι εδώ και η Νίκολα. Ε, δεν ξέρω αν θέλει κάποιος να κάνει ερωτήσεις. Εγώ έχω μια πρώτη ερώτηση και μετά μπορούν να λάβουν το λόγο και οι συνάδελφοι, η οποία αφορά τους πόρους. Διότι τα στοιχεία τα οποία που μας δώσει θα είναι εντυπωσιακά. Τα μισά περίπου από τα παιδιά που γεννιούνται στον κόσμο θα είναι ε, παιδιά από την Αφρική και για την Ιγυρία είναι τα πιο ε, εντυπωσιακά. Μόνο 13 ε, παιδιά στα 100 θα είναι από την Ιγυρία, Χρειαζόμαστε λοιπόν δασκάλους, χρειαζόμαστε κοινωνικούς λειτουργούς κλπ. Πρέπει να επενδύσουμε για την Αφρική λοιπόν, γιατί χωρίς χρήματα, χωρίς χρηματοδότηση, τίποτα από όλα αυτά δεν θα μπορέσουν να υλοποιηθούν. Ε, όταν θα επιστρέψετε, αναφερθήκατε λίγο στη Ρουάντα, μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια μοντέλα ε, που δίνουν τα καλύτερα αποτελέσματα για τα παιδιά. Αντί να επαναλαμβάνετε στοιχεία και αριθμούς, ε, είναι πράγματα με τα οποία ο κόσμος είναι κάπως εξοικειωμένος. Γνωρίζουμε ποιες είναι οι προκλήσεις, αλλά θα θέλαμε να μας πείτε αυτά παραδείγματα. Σε αυτή την περίπτωση λειτουργεί αυτό, για την παιδεία αυτό είναι το καλύτερο μοντέλο, ε, για την πείνα αυτό είναι το καλύτερο μοντέλο, ώστε να μπορέσουμε να αντλήσουμε και κάτω διδάγματα. <coughs> Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. μας ε, παρουσιάσετε μια γενική εικόνα των εξελίξεων στις διάφορες χώρες. Και διαπιστώνται και μεγάλη πρόοδο τα τελευταία 15 χρόνια. Νομίζω ότι αυτά έχουν σχέση και με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης από το 2000 έως το 2015, αλλά και την αξιολόγηση. Κάθε χώρα είχε τα μέτρα της και τα αντίστοιχα αποτελέσματα και βλέπουμε πώς θα πήγαν οι διάφορες χώρες, ποιες πήγαν καλά και ποιες έχασαν αυτή την ευκαιρία. Όσον αφορά τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, ε, υποστηρίζω τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά διαπιστώνω ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων στους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης δεν είναι τόσο σαφής όσο ήταν ε, για τους στόχους της χιλιετίας. Θεωρείτε ότι το βλέπω υπό το σωστό πρίσμα. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε καλύτερη αξιολόγηση και να επιλύσουμε το πρόβλημα, διότι με καλύτερη αξιολόγηση μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να μπορέσουμε να πιέσουμε περισσότερο τις κυβερνήσεις για να δεσμευθούν ε, ακόμα περισσότερο. Και το άλλο έχει σχέση και με αυτό που είπε η Λίντα πώς μπορούμε να αντλήσουμε διδάγματα από κάποιες χώρες ε, που είχαν τις καλύτερες πρακτικές για να έχουμε μεγαλύτερη δέσμευση και καλύτερη και περισσότερη εκπαίδευση. Θα ακούσουμε τις ερωτήσεις και μετά ε, θα ακούσουμε τις απαντήσεις μάλλον ερωτήσεις και μετά θα επανέλθουμε. Ευχαριστώ. Γνωρίζουμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι το μέγεθος των επενδύσεων είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ε, το μοντέλο που προτείνεται για τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης είναι ότι πρέπει να συμβάλλει ο καθένας. Δηλαδή, ε, η κυβέρνηση της κάθε χώρας σε αυτή την περίπτωση είναι η πρώτη η οποία θα πρέπει να συμβάλλει. Και αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι καταρχάς πολλές αφρικανικές χώρες έχουν πόρους και η Νιγηρία. Ορισμένες φορές είναι θέμα διακυβέρνησης, ε, ορισμένες φορές είναι θέμα ε, συλλογής φόρων, ε, διαχείρισης των δημοσίων οικονομικών, αλλά υπάρχουν πόροι σε αρκετές από αυτές τις χώρες. Αυτό που είχε ενδιαφέρον είναι στην έκθεση ότι ακόμα και μια χώρα όπως ο Νίγηρας, που είναι μια από τις 10 φτωχότερες χώρες του κόσμου, μπορεί να κάνει ουσιαστική ε, πρόοδο στον τομέα της εκπαίδευσης, επειδή η κυβέρνηση του Νίγηρα επικέντρωσε τις προσπάθειές της και επένδυσε 22% του προπολογισμού της στην παιδεία. Δεν πιστεύω λοιπόν ότι είναι αδύνατον εάν συνεργαστούν οι εταίροι και οι κυβερνήσεις της Αφρικής, οι χορηγοί, ε, οι εταίροι και ο ιδιωτικός κλάδος επίσης. Ε, νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες στην Αφρική για τον ιδιωτικό τομέα για να μπορέσει και να ε, αποκομίσει κέρδος αλλά να ε, μπορέσει να συμβάλλει και με καινοτομίες ε, στις χώρες στις οποίες θα επενδύσει. Για παράδειγμα, στη Ρουάντα έχουμε ένα παράδειγμα για προϊόντα τα οποία παραδίδονται με drone, κάτι το οποίο δεν γίνεται στην Ευρώπη και είναι κάτι το οποίο συμφωνήθηκε με την Γκάβη ε, για τα εμβόλια τα οποία παραδίδονται μέσω ε, drone και αυτό συμβαίνει όταν έχουμε ανθρώπους από διάφορες περιοχές, ε, τους, ζητούμε, τους βάζουμε γύρω από ένα τραπέζι και τους ζητούμε να λύσουν ένα πρόβλημα. Είναι λοιπόν δυνατό, αλλά απαιτεί ισχυρή πολιτική βούληση και συνέπεια. Δεν μπορεί να αλλάζει κάθε δύο, τρία ή τέσσερα χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι δυνατόν και η Ασία μας δίνει παραδείγματα. Ε, πριν από 15-17 χρόνια ήμουν στην Ινδία, ζούσα εκεί και ε, γεννιόντουσαν 40 εκατομμύρια παιδιά κάθε χρόνο στην Ινδία και σκεφτόμουν πώς θα επιλύσει αυτό το θέμα η Ινδία, διότι πρέπει να συνεχίσουν να χτίζουν σχολεία και κέντρα υγείας, αλλά τα κατάφεραν και προόδευσαν. Υπάρχει λοιπόν κάποια δυνατότητα να γίνουν όλα αυτά. Πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε κάποιες καλές πρακτικές, να γνωρίζουμε βέβαια ότι δεν μπορούμε να αντιγράψουμε τις πρακτικές από τη μια χώρα στην άλλη αυτούσιες, αλλά μπορούμε να δίνουμε τις πρακτικές μας. Υπάρχει και τριγωνική συνεργασία, χώρες όπω η Βραζιλία για παράδειγμα, οι οποίες μοιράζονται πληροφορίες και τεχνογνωσία και πυρογνωμοσύνη με χώρες όπως η Μοζαμβίκη. Υπάρχει δηλαδή ανταλλαγή εμπειριών αυτή τη στιγμή της εξέλιξη. Και κάτι τελευταίο για τις επενδύσεις. Δεν είναι τόσο η ποσότητα των χρημάτων, αλλά η ποιότητα των χρημάτων που επενδύονται. Αν επενδύσουμε περισσότερους πόρους στην εκπαίδευση, αλλά επικεντρωθούμε μόνο στην ανώτατη εκπαίδευση, ε, πανεπιστημιακού επίπεδου, τότε θα έχουμε λίγους καλύτερους ε, φοιτητές οι οποίοι θα παίρνουν πτυχίο, αλλά θα υπάρχει όμως και ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που θα είναι αναλφάβητοι. Ε, και νομίζω ότι δεν υπάρχει ούτε μία αναπτυγμένη χώρα σε αυτόν τον κόσμο που δεν έκανε πρώτα επενδύσεις σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση και μετά. Πρέπει να ξεκινήσουμε λοιπόν από τη βάση. Ε, όσον αφορά τις αξιολογήσεις λοιπά, Εμείς συμφωνούμε, για μας να αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Οι κυβερνήσεις υποτίθεται ότι θα μεταφράσουν τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης σε εθνικούς στόχους και προσπαθούμε να τους βοηθήσουμε να καθορίσουν τις βάσεις για όλα αυτά και μετά από εκεί και πέρα να υπάρχει παρακολούθηση και αξιολόγηση. Και πολλές φορές κάνουμε κοινή αξιολόγηση με τις χώρες ώστε η ποιότητα και ανεξαρτησία των δεδομένων να είναι εγγυημένα. Για παράδειγμα, μια επένδυση στην οποία δύσκολα μπορεί κάποιος ε, να πείσει ότι πρέπει να γίνει με εθνικού πόρους και εδώ νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν και οι εταίροι και οι χορηγοί με τεχνογνωσία και πόρους για να γίνουν αυτές οι αξιολογήσεις, είναι ακριβώς το θέμα των αξιολογήσεων. Και ε, εμείς όμως έχουμε πει ότι πρέπει να ε, μετράτε αυτό το οποίο κάνετε και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Ευχαριστώ. Ο Σάρλ Γκέρεντς θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ και εγώ για την παρουσίασή σας, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και διδακτική. Και αναφερθήκατε στην ανάγκη να είναι οριζόντιες οι διάφορες παρεμβάσεις και μας δώσετε και πολύ συγκεκριμένα παραδείγματα. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Όταν αναφέρεστε στην εκπαίδευση ως τρόπο να περιορίσουμε τον αριθμό των παιδιών ε, αναοικογένεια ή γυναίκα, γιατί ε, αφήνεται στην άκρη τον οικογενειακό προγραμματισμό. Είναι θέμα ταμπού, ξέρουμε ότι είναι λεπτό το ζήτημα, αλλά ακόμα και ο Πάπας είπε ότι ε, δύο παιδιά αναγυναίκα θα έπρεπε να είναι αρκετά. Υπάρχουν λοιπόν στεναρές αντιστάσεις, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αναφέρουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεύτερο, αναφερθήκατε στους παιδικούς γάμους. Ε, εμείς ε, τώρα ξεκινάμε στη διαπραγμάτευση μιας νέας συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρών ΑΚΕ. Νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει και η ερωσιμότητα σε μια τόσο σημαντική συμφωνία βεβαίως. Θα συμφωνούσατε εσείς ή θα προτείνατε στους διαπραγματευτές να είναι μεταξύ των όρων και η απαγόρευση των παιδικών γάμων δύο πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. σε ό,τι αφορά τον οικογενειακό προγραμματισμό δεν είναι θέμα ταμπού σε καμία περίπτωση και η έκθεση το πραγματεύεται. Δεν μπορώ να καλύψω βέβαια όλε τι πτυχέ αυτή τη έκθεση γιατί θα πάρει πολύ χρόνο. Και έχω καταλάβει ότι σα έδωσε ήδη πάρα πολλά νούμερα στην παρουσίασή μου. Στην Αφρική το ποσοστό γυναικών που πραγματικά χρειάζονται τον γενικό προγραμματισμό είναι μεγάλο, 26% σε σχέση με ποσοστά που κυμαίνονται μεταξύ 10-15% στον υπόλοιπο κόσμο. Κάτι που σημαίνει ότι εδώ πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Δεν είναι εντολή της UNICEF, την εντολή την ορίζει Γενική Συνέλευση όπως γνωρίζετε, είναι εντολή του UNFPA, του Ταμείου για τον Πληθυσμό. Και επομένως συνεργαζόμαστε με το UNFPA επιτόπου αλλά και πάλι πράγματι είναι αναλληλένετα τα θέματα, γιατί μιλήσατε και για τη διατομιακή προσέγγιση. Να αναπτύσσουμε γενικέ υπηρεσίες για τα παιδιά, για χωριστά, για τις γυναίκες, για τους άνδρες κτλ. Όχι. Όταν πας σε ένα χωριό, ένα κέντρο υγείας πρέπει να υπάρχει. Και αυτό θα πρέπει να παρέχει ένα πακέτο υπηρεσιών για τον όλο πληθυσμό, για την ε, τοπική κοινωνία και ο γενικό προγραμματισμό πρέπει να εντάσσεται στι υπηρεσίε αυτέ. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι όταν οι γυναίκε ε, μείνουν έγκυε, και πάνε στις ε, υπηρεσίες ε, τις ειδικέ και αν εκεί υπάρχουν εξειδικευμένοι εργαζόμενοι γίνεται μια συζήτηση για το πόσο χρόνο πρέπει να περάσει μέχρι την επόμενη εγκυμοσύνη, αν θα πρέπει να αναβληθεί, να θα πρέπει να διακοπεί κτλ. Πάντως υπάρχει ένα σημείο ε, στο, σύστημα υγείας. Ένα άλλο ενδιαφέρον ήταν ο κόσμος μετά την πολιομήλικτα. Το έχουμε πει και ξανά πολλές φορές, όμως θεωρούμε ότι θα εκριζωθεί τα επόμενα χρόνια η πολιομιλητιδά. Τι κάνει είναι το ερώτημα με τις ομάδες αυτές για την πολιομιλητιδά που είναι επιτόπου παρούσες και δραστηριοποιείται ιδίως σε χώρες όπου το σύστημα υγείας ε, είναι φτωχό και αδύναμο. Με τους εταίρους μας τώρα προσπαθούμε να δούμε πώς ε, θα διαμορφώσουμε διαφορετικά τις ε, μονάδες αυτές ε, που να γίνουν, αν θέλετε, τη σπονδυλική στήλη ενό νέου συστήματο υγεία για τι χώρε αυτέ, ώστε να μην χαθούν αυτοί οι άνθρωποι που έχουν ε, κίνητρα, ε, που είναι ενθουσιασμένοι, με το, μάλλον που είναι στον τομέα αυτό και υπάρχουν πολλέ ευκαιρίε. Θα πρέπει να σκεφτούμε δημιουργικά από εδώ και πέρα. Για να είναι ένα όρο η απαγόρευση των παιδικών γάμων που είπατε. Η συζήτηση είναι μεν ενδιαφέρουσα, αλλά μακάρι να ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, για να το πω έτσι. Σημαντικό είναι γιατί θα στείλει ένα χειρό μήνυμα στον πληθυσμό. Όμως, δεν αρκεί αυτό. Μπορεί κανείς να απαγορεύσει τα ναρκωτικά, μπορεί να απαγορεύσει τη βία σε βάρος των γυναικών και των παιδιών, αλλά και πάλι θα συνεχίσουν αυτά τα φαινόμενα να παρατηρούνται. Το πιο ενδιαφέρον λοιπόν καλύτερα είναι να έχουμε ένα διάλογο με τις κυβερνήσεις για να μας δώσουν να καταλάβουμε τι θέλουν να κάνουν για να σταματήσουν τους παιδικούς γάμους. Είναι πιο πολύπλοκο το καταλαβαίνω, αλλά μια τέτοια συζήτηση θα μπορούσε να γίνει. Και να ενταχθεί και στις απαιτήσει για την παροχή βοήθειας. Τώρα παίρνουμε από την ΤΕΦΚΟ βοήθεια παίρνουμε χρηματοδότηση για να σταματήσουν ε, οι παιδικοί γάμοι και οι ακροτηρισμοί των γυναικείων γεννητικών οργάνων ε, και έχουμε παρουσία, αν θυμάμαι καλά, σε 15 χώρε. Είδαμε ότι ήδη οι κυβερνήσει ενέκριναν από τις 15 νομίζω, οι 12 έχουν ήδη οθετήσει ένα σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση αυτών των δύο ζητημάτων. Και από τις 12 κυβερνήσεις αυτές οι τρεις έχουν ήδη κρίνει ένα προπολογισμό Νομίζω ότι αυτό είναι μια πιο ενδιαφέρουσα πτυχή τη δέσμευση. ότι μια χώρα το παίρνει σοβαρά ε, όταν έχει ένα νόμο ή όταν έχει ένα σχέδιο. Αν το βάλουμε προϋπόθεση, όρο, ίσω και δεν θα το κάνουν. Δεν θα βελτιωθεί δηλαδή κατά ανάγκη και η ζωή των παιδιών επιτόπου. Με τη UNICEF, το UNFPA και την κοινωνία των πολιτών νομίζουμε ότι η προσέγγιση αυτή και η συζήτηση αυτή είναι πιο ενδιαφέρουσα και θα μπορούσε να οδηγήσει και σε πιο απτά αποτελέσματα. Πρόεδρος. Φαντάζομαι ότι σε πολλές χώρες είναι παράνομο, μεν, αλλά συμβαίνει. Είναι παραδοσιακό, ε, παραδοσιακές πρακτικές όπως ο κρατασμός για των γενικών οργάνων παρά την νομοθεσία και την καλή διακυβέρνηση. Δεν βλέπω να θέλει κάποιος άλλος να έρθει στο λόγο. Όμως έχουμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Φαμπιέν Βαντενάιτ και τον Ιθ, τον κύριο Εκμεζόγλου, κάπω έτσι. Δυστυχώ δεν μπορώ να προφέρω σωστά τον. Από τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ παρακαλώ, το λόγο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα ήθελα να σα ευχαριστήσω για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Καλωσορίζουμε τη μελέτη αυτή. Κοιτώντα ε, τη σύνοψη και τα αποτελέσματα, θέλω να υπογραμμίσω ότι είναι ύψη τη σημασία η επένδυση στα παιδιά όπως πολύ σωστά είπατε, αποτελεί βασικό στόχο μεταξύ των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπου τα αγόρια και τα κορίτσια παίζουν σημαντικό ρόλο. Ήθελα επίσης να υπογραμμίσω πόσο μεγάλη σπουδαιότητα δίνεται σε όλα τα παιδιά στη νέα συνένεση για την ανάπτυξη που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου και η νεολαία αποτελεί οριζόντιο ζήτημα. Μετά από αυτή τη συνένεση έχουμε προγραμματίσει διάφορα έργα, διάφορα προγράμματα όπως ε, το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο που ενθαρρύνει επενδύσεις στην Αφρική που εξετάζει τα έθραυστα περιβάλλοντα. Έχουμε την πρωτοβουλία Αφρικανικής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ξεκινήσει νομίζω για την εξέλιξη της βίας κατά των γυναικών Πρόκειται για ένα έργο το οποίο υπάρχει εδώ και καιρό, αλλά θα εστιαστεί ιδιαίτερα στην Αφρική αυτή τη στιγμή. Έχουμε διάφορα έργα τόσο για τα επιστοποιητικά γέννηση, για τα ισπαιδικού γάμου. Και όπω είπε και η πρόεδρο, έχουμε την επερχόμενη Σύνοδο Κορυφή Αφρικανική Ένωση και Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε και άλλα προγράμματα ε, για διάφορους τομείς όπως η παιδεία. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης θέλετε να πείτε κάτι. Ναι, με ακούτε. Εγώ είμαι η κυρία με το δύσκολο όνομα, η κυρία Εκμετζόγλου. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα για να συμπληρώσω την Επιτροπή η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ε, συνομιλεί τακτικά με τη UNICEF. Είχαμε και την ευχαρίστηση να δεχθούμε και περιφερειακού διευθυντέ τη Αφρική που μα παρουσίασαν διάφορε μελέτε. Ε, παρακολουθούμε λοιπόν πολύ στενά την ιδρυτική σχέση με τη UNICEF. Όσον αφορά του στόχου βιώσιμη ανάπτυξη από του συναδέλφου σα και από οι δικοί μου συνάδελφοι εδώ, του στόχου αυτού πρέπει να του βλέπουμε στο σύνολό του ω οριζόντιο, ω εγκάρσιο θέμα, ω θεματολόγιο το οποίο θα πρέπει να μας απασχολεί στο σύνολό του. Το θέμα λοιπόν των παιδιών θα πρέπει λοιπόν να δοθεί στο πλαίσιο καθενός από τους στόχου βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο πρέπει να στείλουμε. Και συνεργαζόμαστε με την Κομισιόν μέσω διαφόρων έργων όπως προαναφέρθηκε για να αξιοποιήσουμε αυτά, τον αλληλένδετο χαρακτήρα των διαφορών θεμάτων. Δεν υπάρχει λοιπόν μία λύση, πρέπει να ε, σπάσουμε τα στεγανά. Όπως είπαμε στη Σύνοδο αυτή κορυφή θα συζητηθεί το ζήτημα της νεολαίας και συνεργαζόμαστε στενά για την προετοιμασία με την Αφρικανική Ένωση. Η νεολαία πιστεύω είναι αυτή που μας απασχολεί περισσότερο ο ζήτημα στο σύνολό της. Ευχαριστούμε πολύ και για την παρουσίαση και για τη μελέτη. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Ε, αυτό που είπε ο Τσάρλς για τις γυναίκες, ε, υπάρχει και μελέτη EPRS, ε, αυτό που ονομάζεται παγκόσμιος, παγκόσμιος μετρητής τάσεων που εξετάζει τα δημογραφικά στοιχεία και λέει ότι το όλο δημογραφικό ζήτημα αφορά τη χειραφέτηση των γυναικών, την εκπαίδευσή του, ε, τι επιλογέ που κάνουν οι γυναίκε εφόσον έχουν χειραφετηθεί και εφόσον έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτέ τι ε, επιλογέ. Κοιτάζω τώρα το Ροσάριο για την γραμματεία. Μπορείτε να στείλετε ε, ένα link στου συναδέλφου για να μπορούν να βρουν αυτή τη μελέτη. Διότι πιστεύω το ζήτημα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν κλείσουμε. Θέλω να πω ότι πράγματι πιστεύω ότι όλα τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Η δική σας επιτροπή, υπερθυμίζοντας την Ένωση ότι για αναπτυξιακή βοήθεια θα πρέπει να συνεχίσει να εστιάζει την ανάπτυξη. Αλλά θα πρέπει να γίνουν σημαντικές επενδύσεις. Αυτό δεν μπορεί να παρακαμφθεί και να αγνοηθεί. Η μετανάστευση δεν τα καλύψει όλα και χαίρομαι που κανείς δεν μίλησε για τη μετανάστευση. Ίσως είναι η πρώτη φορά από τότε που έρχομαι εδώ που κανείς δεν με ρώτησε για μετανάστευση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στα θεμελιώδη στοιχεία της ανάπτυξης για τις αυσκανικές χώρες και σε άλλες χώρες βέβαια του κόσμου. Τα παιδιά συχνά τα παραβλέπουμε επειδή δεν ψηφίζουν, δεν κατεβαίνουν στους δρόμους να διαδηλώσουν, ωστόσο γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει καμιά χώρα στον κόσμο που να πέτυχε και να ανεπτύχθη χωρίς να έχει επενδύσει τα παιδιά στην υγεία τους, στην παιδεία τους, στην προστασία τους. Και νομίζω ότι εδώ η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι απλά μπορεί να υποστηρίξει με χρηματοδότηση, αλλά και με τη φωνή της. Γιατί έχετε τις ίδιες αξίες. Αναφέρεστε στη συνθήκη της Λισαβόνα στα δικαιώματα των παιδιών. Επομένω, η εταιρική σχέση για τα παιδιά θα πρέπει να προχωρήσει σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις, ε, την παροχή βοήθειας και τεχνογνωσίας, εμπειρίας. Σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε. Ήταν πάρα πολύ ε, σημαντικό, ιδίω τη μέρα αυτή που είναι αφιερωμένη στα παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαστε πάντως στη διάθεσή σας αν έχετε περισσότερες απορίες. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Είπα και σήμερα ότι ξεκινήσαμε τα παιδιά, έχουμε διάφορα στήματα, θα μιλήσουμε μετά για την Αφρικανική στρατηγική και μετά για τις επενδύσεις. Γιατί είναι, έχουμε ένα θέμα, έτσι, μια θεματολογία αυτή την εβδομάδα. Και με τα παιδιά νομίζω κάναμε την καλύτερη δυνατή αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι, αλλάζει το πάνελ. Θα έχουμε μια αξιολόγηση της κοινής στρατηγικής Ευρωπαϊκής Αφρικής για να αλλάξει λίγο το πάνελ, δύο λεπτά διάλειμμα. Okay, colleagues, we now move on to item Αγαπητοί συνάδελφοι, να περάσουμε τώρα στο σημείο 6, μια παρουσίαση μελέτης που εκπώνησε για την Επιτροπή μας και το Αφρικαϊκό Κοινοβούλιο. Επειδή έχουμε και τη διάσκεψη μόνη εβδομάδα στα Μπιτζάν, Για τη στρατηγική λοιπόν, κατά πόσο είστε με επιτυχία μέχρι τώρα, το 2007 εγκρίθηκε στρατηγική και διέπει τη σχέση με αυτή, Υπήρξαν διάφοροι οδικοί χάρτε. Και ελπίζουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα να εγκριθεί μια διακήρυξη στο Αμπιτζά. Από το 7 έχουν αλλάξει πολλά, έχει αλλάξει ο κόσμος. Έχουμε τους στόχους ε, της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, με τους στόχους της και περιμένουμε να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, νέες προκλήσεις, τη γονιμότητα, τη δημοκρατία. Θέλουμε να ακούσουμε λοιπόν από εσά μια ανάλυση για το τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και για το τι θα μπορούσε να ακολουθήσει να συμβεί και στο μέλλον. ξεκινήσουμε με την Νικόλα που είναι επικεφαλή του προγράμματο για το European International Relations Manager. Κύριε Πυρότση, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι πολύ και εγώ και οι συναδελφοί που είμαστε εδώ να σας παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης που διεξήγαμε για την κοινή στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης 10 χρόνια μετά, κριτική εξέλιξη και προοπτικές. Πρώτα απ' όλα τι κάνει αυτή η έκθεση αξιολογεί την ε, υλοποίηση πρώτα απ' όλα της εκείνης στρατηγικής, ιδίως στον οδικό χάρτη 2014-2017, που ήταν ε, το τελευταίο έγγραφο υλοποίησης μέχρι στιγμής, ότι τη στρατηγική. Δεύτερον, αξιολογεί τις προτεραιότητες που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόσφατη κοινή ε, ανακοίνωση για μια νέα όθηση στην εταιρική σχέση Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος ε, παρέχει συστάσεις για ενισχυμένη συνεργασία Αφρικανικής Ένωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, εν ώψη και της προσεχούς διάσκεψης κορυφής στο Αμπιτζάν, στα τέλη Νοεμβρίου. Στην παρουσίασή μας, έχω με νομίζω 20 λεπτά λίγο πολύ στη θέση μα, θα ήθελα λοιπόν να σα παρουσιάσω πρώτα απ' όλα τα γενικά πορίσματα σε ό,τι αφορά τη μέχρι τώρα υλοποίηση της κοινή στρατηγικής και έπειτα θα σας παρουσιάσουμε τις συστάσεις που θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικές ε, για την ε, πολιτική που ακολουθεί η Ένωση και τα θεσμικά της όλων. Πρώτα απ' όλα, σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση της υλοποίησης της κοινή στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής 10 χρόνια λοιπόν, αφού το εγκρίθηκε το 2007, βρήκαμε ότι οι βασικές προτεραιότητες που ορίστηκαν το 2007 σε αυτήν την εταιρική σχέση εξακολουθούν να ισχύουν. Ωστόσο θα πρέπει να επικαιροποιηθούν για να λάβουν υπόψη το μεταβαλλόμενο πλαίσιο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στην Αφρικανική Ήπειρο και το μεταβαλλόμενο διεθνές πλαίσιο εν γέννη. Και ιδίω σε σχέση με τα δύο βασικά στρατηγικά έγγραφα που εγκρίθηκαν πρόσφατα από την Αφρικανική Ένωση και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τη μία την Ατζέντα 2063, το θεματολόγιο που ουσιαστικά ε, αναφέρει ποιος πρέπει να είναι ορίζοντας για τις αλλαγές, τις κοινωνικές αλλαγές για τα επόμενα 50 χρόνια στην Αφρική. Και έχουμε την Παγκόσμια Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα στρατηγικό έγγραφο που αναμορφώνει ε, την ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ε, τη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επόμενα χρόνια ποιοι είναι οι προεξέρχοντες στόχοι της ήδη εταιρικής σχέσης. Βλέπουμε ότι οι πολιτικές πτυχές ε, ήταν αντικείμενο ένας πολυεπίπεδου συστήματος με διασκέψεις που γίνονταν στην Ευρώπη και στην Αφρική. Όμως αυτός ο πολιτικός διάλογος υψηλού επίπεδου δεν ε, είναι επαρκής ιδίω σε υπουργικό επίπεδο, πρέπει να ενισχυθεί λοιπόν στο μέλλον. Υπήρξαν βέβαια πρόσφατα επιθέσεις της ε, προσώπα του Προέτσης Κομισιόν και είναι ένα σωστό βήμα αυτό, αλλά πρέπει να γίνουν και άλλα. Δεύτερον, οι κλιματοοικονομικές πτυχές. Σημαντικός, κρίσιμος παράγοντας των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικανικής Ένωσης. Θεωρήσαμε πάντω ότι είναι πολλά τα δημοσιονομικά προγράμματα, τα χρηματοοικονομικά προγράμματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει και μεγάλη εξάρτηση από την άλλη πλευρά των Αφρικανών εταίρων από τη χρηματοδότηση που έρχεται από εξωτερικό και ιδίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, παρά το ότι ο στόχος ε, της εταιρική σχέση αρχικά ήταν ανθρωποκεντρική και να δημιουργήσει μια πιο ισορροπημένη σχέση μεταξύ των ε, δύο πλευρών, είδαμε ότι παρά τις εκκλήσεις ε, δεν συμμετέχουν αρκετά, για παράδειγμα, οι οργανώσεις και των πολιτών σε αυτή την εταιρική σχέση. Παραμένει δηλαδή μη ισορροπημένη. Εδώ ε, περιορίστηκα λοιπόν σε κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Αν ε, δείτε και το τελευταίο εγγραφό που αναφέρει ποιες είναι οι προτεραιότητες για την κοινή στρατηγική που ήταν ο δικός χάρτης 2014-2017 τα αποτελέσματα είναι μεικτά σε ό,τι αφορά την υλοποίηση. Η μεγαλύτερη έλλειψη, η μεγαλύτερη αδυναμία της εταιρικής σχέσης είναι ότι δεν έχει ε, ενεργοποιήσει τον πολιτικό διάλογο στο ύψιστο επίπεδο. Ιδίως για τα πιο επίμαχα ζητήματα, όπως είναι για παράδειγμα μετανάστευση, διεθνής δικαιοσύνη, ανθρώπινα δικαιώματα και μεταρρύθμιση της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Μια άλλη αποτυχία είναι ε, το ετήσιο φόρουμ, το κοινό ετήσιο φόρουμ, όπου δηλαδή οι ιδιωτικοί τομεί ε, και οι κοινωνίε ε, και οι οργανώσει πολιτών από τι δύο πλευρέ θα αξιολογούσαν τη στρατηγική και θα κατέθεταν προτάσει. Αυτό είναι ένα από τα βασικά κενά που πρέπει να καλυφθεί. Καλύψαμε τώρα τρεις βασικούς τομείς. Η ειρήνη και η ασφάλεια. Συνεργασία για τη δημοκρατία και η χρηστή διακυβέρνηση και Προώθηση επενδύσεων και επιχειρηματικότητα. Σε ό,τι αφορά το πρώτο, ειρήνη και ασφάλεια. Είναι αδιαφυσβήτητο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει πολύ σημαντικό εταίρο τη Αφρικανική Ένωση και σε ό,τι αφορά την τεχνική υποστήριξη και σε ό,τι αφορά τη χρηματοοικονομική υποστήριξη. Όμω υπάρχουν, όπω είπα, προβλήματα που έχουν να κάνουν με την πολυπλοκότητα και τον κατακαιρματισμό των χρηματοδοτικών προγραμμάτων. Και δεν υπάρχει επαρκή απορροφητικότητα των κονδυλίων. Υπάρχουν όμως προγράμματα ενδυνάμωσης και καθοδήγησης που ε, δεν έχουν ακόμη φέρει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα γιατί υπάρχει εξάρτηση των, της αφρικανικής πλευράς από το εξωτερικό. Σε ό,τι αφορά τη διακυβέρνηση πολλά μπορούν να γίνουν και τη δημοκρατία. Ιδίω ό,τι αφορά την υποστήριξη της αρχιτεκτονικής της διακυβέρνησης θα πρέπει να ε, υπάρξει υποστήριξη μεγαλύτερη και να εστιάσουν πιο πολύ δύο πλευρές στα πρακτικά ζητήματα. Στο τρίτο θέμα τώρα υπάρχει κάποια σύγχυση. Μέχρι στιγμής. Μείωση φτώχεια, εκδημοκρατισμό, δημιουργία θέσεων, εργασία είναι οι στόχοι του οδικού χάρτη. Δεν αρκούν. Δεν υπάρχει ένα συνεκτικό πλαίσιο συνεργασία για τα σημαντικά αυτά ζητήματα μέχρι τώρα. Περνάμε στι συστάσει τώρα προείπα ότι σε γενικό επίπεδο αυτό που θέλαμε ήταν να υπογραμμίσουμε την ανάγκη πρώτα απ' όλα να υπάρξει ένας βελτιωμένος, ενισχυμένος πολιτικός διάλογος με πιο συχνές επαφές σε υπουργικό επίπεδο μεταξύ δηλαδή των Υπουργείων Αφρικανικής Υπήρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χρειάζεται ένας χρειάζεται μια ενίσχυση και μια υποστήριξη από τι εθνικέ κυβερνήσει, αλλιώ δεν πρόκειται να βελτιωθούν οι σχέσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση Αφρική στον τομέα τη ειρήνη και τη ασφάλεια. Είναι σημαντικό να ενισχυθεί ο διάλογο μεταξύ ε, του Συμβουλίου Ειρήνη και Ασφάλεια ε, του τη Αφρικανική Ένωση και τη αντίστοιχη επιτροπή ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην μείνετε μόνο στην ανταλλαγή πληροφοριών και να είναι πιο συχνέ οι επαφέ μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Παναφρικανικού Κοινοβουλίου αλλά και Αφρικανικών Κοινοβουλίων σε εθνικό επίπεδο, σε ό,τι αφορά ε, χρηματοδοτικούς μηχανισμούς και προγράμματα. Πρέπει πρώτα απ' όλα να μειωθούν οι πρωτοβουλίες και να είναι και πιο συνεπείς, συνεκτικές μεταξύ τους. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το 2014 που καλύπτει αποκλειστικά τη, τα χρηματοδοτικά προγράμματα για την υλοποίηση της κοινή στρατηγική σε Αφρικανικό επίπεδο. Δεν είναι όμως αρκετή η χρηματοδότηση και δεν υπάρχει και επαρκής διασύνδεση με άλλα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάντα από πλευρά της, Ευρωπαϊκ... της Αφρικανικής Ένωσης πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ε, κινητοποίηση πόρων χρηματοδότηση και σε ό,τι αφορά την αμοιβαιότητα, ιδίως στον τομέα της παιδείας και της ε, εκπαίδευσης κατάρτισης. Πρέπει να υπάρχουν περισσότερες ανταλλαγές και σε τοπικό επίπεδο. Πρέπει να είναι προτεραιότητα για το άμεσο μέλλον. Και θα ολοκληρώσω τη δική μου παρέμβαση με μια συγκεκριμένη σύσταση ότι αφορά την ειρήνη και ασφάλεια, που είναι μια από τι βασικέ προτεραιότητε τη κοινή στρατηγική και μια από τι βασικέ στρατηγικέ και στον πιο πρόσφατο οδικό χάρτη. Ένα από του βασικού στόχου εδώ είναι η αρχιτεκτονική ειρήνης και ασφάλειας και η stand-by force, ε, η δύναμη αυτή εφέδρων, θα πρέπει να γίνουν επιχειρησιακά αυτά τα δύο. Γιατί εδώ έχουμε πρόβλημα, υπάρχει καθυστέρηση. Πρέπει να επαναξισορροπηθεί η χρηματοδότηση που δίνεται για τις ειρηνευτικές επιχειρήσεις υπέρ της δημιουργίας υποδομών ε, και θεσμών στην ε, Αφρικανική Ήπειρο. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο και για πρόοδο και για να πολλαπλασιαστούν οι προσπάθειες ώστε να συνεισφέρει περισσότερο στο Ειρηνευτικό Ταμείο η Αφρική, που και το βασικό εργαλείο που υπάρχει ε, για να δοθεί ε, πραγματικά αφρικανική λύση στο πρόβλημα και να ειδοποιηθούν οι Αφρικανοί αυτή την προσπάθεια. 0,2% είναι ένας φόρος μιας φορά που έχει προταθεί ε, για τις αφρικανικές χώρες που θα χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της Αφρικανικής Ένωσης και του Ειρνευτικού Ταμείου. Δεν έχει ξεκινήσει να συλλέγεται τη σφορά αυτή. Υπάρχουν λίγες εξαιρέσεις αφρικανικές χώρες και θα σταματήσω εγώ εδώ και θα συνεχίσω την παρουσίαση στην συνάδελφοί μου. Ευχαριστώ. Όσον αφορά τη δημοκρατία, την καλή διακυβέρνηση και τα ανθρώπινα δικαιώματα, το πρώτο το οποίο θα ήθελα να επισημάνω και έχει σχέση με την κοινωνία των πολιτών, είναι πάρα πολύ σημαντικό στο μέλλον να εξασφαλίσουμε πραγματική συμμετοχή παραγόντων της κοινωνίας των πολιτών, πέραν ε, των γενικών ε, τυπικών δηλώσεων. Όπως είπα προηγουμένως, το πρώτο συγκεκριμένο βήμα θα μπορούσε να είναι η σύσταση του ε, κοινού ετήσιου φόρουμ για να συζητήσουν τα πιο επίμαχα ζητήματα μεταξύ Αφρικανών και Ευρωπαίων εταίρων και να επιλέξουν και τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και των ενδιαφερομένων που θα συμμετέχουν. Ένα δεύτερο στοιχείο αφορά την ευρύτερη οπτική της δημοκρατικής διακυβέρνησης και της συμμετοχής των πολιτών σε αυτή την εταιρική σχέση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υποστηρίζει τις εκλογικές διαδικασίες ε, και αυτό ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά η δημοκρατική διακυβέρνηση δεν είναι μόνο οι εκλογές και επομένως οι προσπάθειες θα πρέπει να πηγαίνουν πέραν μιας απλής εκλογικής αναμέτρησης. Για παράδειγμα, ακόμα και ο ρόλος των κοινοβουλίων θα μπορούσε να ενισχυθεί και να αυξηθεί ο ελεγκτικός ρόλος του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή της στρατηγικής. Τρίτον, τα θέματα φύλου θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη με συγκεκριμένα μέτρα ισότητα φύλων και ενδυνάμωση των γυναικών. Όλα αυτά θα πρέπει να τα υποστηρίξουμε μέσω, για παράδειγμα, σύστασης δικτύων μεταξύ Ευρωπαίων και Αφρικανών εταίρων. Αυτό θα μπορούσε να γίνει και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο μεταξύ ε, ε, βουλευτών της Παναφρικανικής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. για τις εξελίξεις ανθρωπιστικά θέματα. Η πρώτη προτεραιότητα που τονίζουμε στην έκθεσή μας αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών. Ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα αναφέρονται σε πολλά έγγραφα βεβαίως, αλλά η εντύπωση που δίνεται είναι ότι δεν υπάρχει κατάλληλος εξορθολογισμός και δεν συμπεριλαμβάνονται σε κάθε συμφωνία μεταξύ Ευρωπαίων και Αφρικανών εταίρων. Επίσης, οι τάσεις ε, ε, μεγαλύτερης ασφάλειας θα πρέπει να περιοριστούν και θα πρέπει ε, να διευκρινιστεί η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης συνόρων. Κατόπιν υπάρχει και μία σύσταση για τη σχέση μεταξύ της ανάπτυξης και της ασφάλειας. Είναι πολύ στενή μεν αυτή η σχέση, αλλά δεν είναι ταυτόσιμη. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε αυτή τη σχέση, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε κατά νου και την ανάπτυξη ως ένα συγκεκριμένο στόχο που θέλει να εκριζώσει την φτώχεια. Η πολιτική ανάπτυξη λοιπόν θα πρέπει να επικεντρώνεται πολύ συγκεκριμένα στο θέμα αυτό και όλες οι πολιτικές θα πρέπει να προσανατολίζονται στις προτεραιότητες των αφρικανικών και ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή την εκρίζωση της φτώχειας και όχι να τα αφιερώνουμε απλώς στον περιορισμό και στην ε, αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών. Είναι σημαντικό και αυτό, αλλά δεν είναι ε, ο πρωταρχικός ρόλος της αναπτυξιακής πολιτικής. Από εκεί και πέρα μας ενδιαφέρουν ε, οι διάβλοι νόμιμης μετανάστευσης. Αυτό θα πρέπει να είναι τμήμα μιας δέσμης μέτρων που θέλει να μειώσει την παράνομη μετανάστευση, να καθορίσει ε, νόμιμους διάβλους που θα σχετίζονται με ευκαιρίες απασχόλησης που είναι ένας από τους τρόπους να έχουμε ένα νόμιμο διάβλο και μια ασφαλή οδό μετανάστευσης χωρίς ε, να υπάρχουν ε, ε, θέματα έλλειψης ασφάλειας και κινδύνου. Και υπάρχει και μία σύσταση που αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες και τον αλφαβητισμό. Πιστεύουμε ότι μαζί με τις ψηφιακές τεχνολογίες ε, θα μπορέσουν να συμβάλλουν σε καλύτερη ε, κοινωνική εξέλιξη που δεν θα αποκλεί κανέναν. Ευχαριστώ Μπερνάρντο. Όσον αφορά τώρα τους τελευταίους δύο τομείς προτεραιότητες ε, ε, αφορούν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Ε, σήμερα, όπως είπε και η Νικολέτα, οι μηχανισμοί που αναφέρονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να βοηθήσουν τις επενδύσεις στην Ήπειρο είναι πολύ περίπλοκοι και πολύ δύσκολο να τους αντιμετωπίσουν οι επενδυτές. Έχουμε τέσσερις συγκεκριμένε συστάσεις, οι οποίες μπορούν να δώσουν μια όθηση σε μια ανάπτυξη που θα είναι βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ε, και ε, κυρίως ε, μας ενδιαφέρει η εκμετάλλευση των πόρων με βιώσιμο τρόπο, ώστε να μπορέσει να υπάρχει κατάλληλη χρήση πόρων στην Αφρική που αποτελούν και πάρα πολύ σημαντικό σκέλος του εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Επίσης, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων πολύ σωστά αναφέρεται και στην κοινή ανακοίνωση για να συμπεριλάβει και κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς ε, παράγοντες. Αλλά η δυσκολία της ε, ε, ανακοίνωσης είναι πώς μπορούμε να αξιολογήσουμε πραγματικά αυτούς τους παράγοντες και να τους εντάξουμε στο διάλογο. Επιπλέον, οι στόχοι της βιωσιμότητας και της περιβαλλοντικής προστασίας θα πρέπει να μπορέσουν να ενταχθούν κατά τρόπον ώστε να επεκτείνουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για τη διαχείριση των φυσικών πόρων. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει ένα παναφρικανικό υποχρεωτικό πλαίσιο για τη διαχείριση των φυσικών πόρων, τουλάχιστον να υπάρχει κοινό έδαφος ώστε να εγγυηθούμε αφενός επαρκέ σε επίπεδο επενδύσεων από το εξωτερικό και ταυτόχρονα να δώσουμε και περισσότερη εξουσία για να ελέγχεται η συμπεριφορά όλων εκείνων που συμμετέχουν σε αυτόν τον συγκεκριμένο τομέα. Εξετάζοντας τους πόρους, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναπτυχθεί και να ε, ε, βοηθήσουμε τις τοπικές δυνατότητες ε, κυρίως προς όφελος των πολιτών της Υπήρου των ε, επιχειρήσεων της Υπήρου και αυτό είναι ο μόνος τρόπος ο οποίος θα δώσει όθηση και θα ενισχύσει την εσωτερική ζήτηση για το αφρικανικό εμπόριο που είναι και ένας από τους στόχους της ίδιας της στρατηγικής. Σήμερα το εμπόριο αγαθών μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής κυρίως βασίζεται σε πρώτες ύλες και φυσικούς πόρους. 50 με 60% αυτών των πόρων φτάνουν στην Ευρωπαϊκή ε, Ήπειρο χωρίς καμία διαδικασία μεταποίησης ε, στο ενδιάμεσο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσουμε τη διαδικασία ανάπτυξης στην Ήπειρο, επομένως να ε, δώσουμε τη δυνατότητα να μεταποιούν οι ίδιοι τους φυσικούς τους πόρους. Για να γίνει αυτό, πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα και στο θέμα της διαχείρισης της ενέργειας και στην πρόσβαση σε εξουσία. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν ε, αξιόπιστα ρυθμιστικά πλαίσια για τους επενδυτές και είναι πάρα πολύ σημαντικό και από πλευράς αφρικανικών λοιπόν θεσμικών οργάνων να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο για να μπορέσουν να ανοίξουν και να προλιάνουν το έδαφο ε, για όλες αυτές τις επενδύσεις. Ταυτόχρονα όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημαντικές δυνατότητες να συνεργαστεί με τους εταίρους της όπως έκανε και στη Μεσόγειο για παράδειγμα με το Ίντερε και το Μέτζο πρωτοβουλίες οι οποίες ε, βοήθησαν τις ρυθμιστικές αρχές στην περιοχή να συνεργαστούν ε, για να μπορέσουν ε, να έχουν βασικά ρυθμιστικά πλαίσια και το MEDREG και το MEDTSO για τους ρυθμιστές συστημάτων μεταφορών για να μπορέσουν να προσδώσουν και συγκεκριμένη δυνατότητα σε επενδυτές. Τέλος, να εκμεταλλευτούμε τα όσα συνέβησαν στον ε, αγροδιατροφικό τομέα, ε, κυρίως όσον αφορά την επισητιστική ασφάλεια και την τεχνολογία που αφορά την επισητιστική ασφάλεια και τη διατροφή, ώστε να μπορέσουμε να μεταλαμπεδεύσουμε και τεχνολογίες δημιουργίας δυνατοτήτων ε, ε, σε αυτό τον τόσο συγκεκριμένο σημαντικό τομέα και διαδικασίες αυτοματισμού επίσης, ε, όλα αυτά τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, διότι ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι να έχουμε τους πολίτες της Αφρικής στο επίκεντρο της διαδικασίας και να τους προσφέρουμε και τα μέσα να προσελκύσουν επενδύσεις για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε από τη βάση το συγκεκριμένο τομέα. Και αυτό φυσικά ε, σημαίνει ότι αυτό θα είναι και προς όφελος ε, του γενικότερου εμπορίου μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής και θα μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να βρούμε και νέους τρόπους ε, να ε, αντικαταστήσουμε τα πλαίσιο του EPA που δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό όσο περιμέναμε. Τέλος, ε, κάποιες προκλήσεις για τις παγκόσμιες ε, προκλήσεις που έχουν, κάποιες συστάσεις για τις παγκόσμιες προκλήσεις είχαμε συστάσει από τις τελευταίες COP από το Παρίσι και μετά ε, να ενισχύσουμε τη σχέση μεταξύ ενεργειακών πολιτικών και δράσης για το κλίμα. Η δράση για το κλίμα είναι θεμελιώδες ε, ζήτημα σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Αφρική και για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπάρχουν διάφορες προκλήσεις οι οποίες ε, τίθενται στις κοινωνίες μας και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει πολύ φιλόδοξες ε, πρωτοβουλίες ε, στη διαδικασία των μετριασμού των συνεπειών, για παράδειγμα χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ε, νέες δυνατότητες για πιο καθαρή ενέργεια, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μπορούσαμε να κάνουμε και κάποια περισσότερα πράγματα όσον αφορά τη διαδικασία της προσαρμογής, διότι δυστυχώς οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής θα πλήξουν της Υπήρους ή την Ήπειρο, επομένως θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και αυτές τις προσα... Ε, προκλήσεις προσαρμογής που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη στρατηγική. Μια ακόμα σημαντική πτυχή είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε και να δώσουμε όθηση για την ε, πράσινη χρηματοδότηση ε, που δεν αφορά μόνο ενεργειακά προγράμματα αλλά και οικονομικό και βιομηχανικό κλάδο της Αφρικανικής Υπήρου. Θα πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ε, ατζέντα ανάπτυξης του 2030. Ε, σήμερα συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής δεν έχει καμία σχέση με τα όσα είχαν καθοριστεί με την ε, πρωτοβουλία της ανάπτυξης της χιλιετίας ε, της Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά θα πρέπει να τα προωθήσουμε ώστε να το συμπεριλάβουμε στην εταιρική σχέση όχι μόνο στα δύο στρατηγικά έγγραφα, να συμπεριλάβουμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης ε, στην ίδια την εταιρική σχέση και κυρίως να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε και σε τοπικό επίπεδο αυτά τα οποία ε, περιλαμβάνονται στους στόχους της ε, βιώσιμης ανάπτυξης. Και τέλος να συζητήσουμε και να θέσουμε τη Σύνοδο Κορυφής ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής σε θέση να συζητήσει διάφορες λύσεις μετά το κοτονού. Εάν τα αποκλείσουμε σημαίνει ότι θα παραβλέψουμε κάποια επίμαχα ζητήματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να τα αφήσουμε ανοιχτά αυτά και να προσδώσουμε αξία και στη σχέση της Αφρικανικής Ένωσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πλαίσιο αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επισκόπηση. Πολύ επικαιρό με τη Συνοδοκορυφή στην επόμενη εβδομάδα. Έχω τον Σάρλα πρώτο που θέλει να μιλήσει. Κύριος Γκέρεντς, ε, έχω πολλές ερωτήσεις. Ε, θα επικεντρωθώ σε κάποια σημεία που θεωρώ πολύ βασικά. Η κυρία ε, Πύροτσι αναφέρατε την εταιρική σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής στο πλαίσιο του πολιτικού διαλόγου και λέτε ότι λυπάστε που δεν γίνονται αρκετές συναντήσεις. Ε, μεταξύ δύο συνόδων κορυφή σε υπουργικό επίπεδο. Πιστεύω ότι όταν μιλάμε για στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για την Αφρική. Είναι σαν να αναρωτιόμαστε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τον κόσμο με μια πολύ πάγια στρατηγική. Ε, για να βελτιώσουμε τον κόσμο πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε εδώ, στα σπίτια μας. Δεν με εκπλήσει που δεν λειτουργεί ο πολιτικός διάλογος. Αν δεν υπάρχουν αρκετοί υπουργοί σε αυτές τις ε, συναντήσεις, τι να γίνει, πρέπει να δείτε πόσοι υπουργοί είναι όταν γίνονται αντίστοιχε σύνοδοι και εδώ. Αν δεν υπάρχουν υπουργοί για να τους στείλουν ε, στο Συμβούλιο Ανάπτυξης, πώς να υπάρχουν υπουργοί για να τους στείλουμε στη... να συζητήσουν την ανάπτυξη στην Αφρική. Και επίσης πρέπει να δούμε κατά πόσο έχουν την εξουσιοδότηση να μιλήσουν εξ ονόματο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θυμάμαι στην Κινσάσα το 2010 νομίζω, κανένας υπουργό δεν υπήρχε που να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στη συνάντηση ε, μικτής ε, κοινοβουλευτικής επιτροπής ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και διότι η κυρία Άστον είχε αποφασίσει έτσι να μην υπάρχει κανένα. Αυτή θα εκπροσωπούσε όλου, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Θα πρέπει να βάλει λίγο τάξη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα αυτά και να αποφασίσει ποιο κάνει τι και με τι εντολή. Δηλαδή πρέπει να οριστούν διάφορες αποστολέ. Εδώ βρισκόμαστε σε μηδενικό σημείο. Δεν αμφιβάλλω ότι η κυρία Μογκερίνη, ναι, είναι ένας ταλαντούχος άνθρωπος, γνωρίζει το αντικείμενό τη, ε, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα. Πρέπει να μάθουμε να αναθέτουμε, να εκχωρούμε αρμοδιότητες και σε άλλους. Ε, οπότε πρέπει να κάνουμε κάποια ενδοσκόπηση, να δούμε λίγο τι γίνεται μεταξύ μα. Το δεύτερο που ήθελα να αναφέρω αφορά την σύσταση που ακούσαμε από τον κύριο Σαρτόρη νομίζω στο τέλος είπε ότι είναι αναγκαίο να δούμε τι γίνεται και μετά ε, Κοτονού, Αμπιτζάν ναι εννοείται θα χρειαστεί κάποιο χρόνο για να έχουμε τέτοια πάνελ προσωπικότητων να αναφέρουν αυτά τα ζητήματα. Το θέμα είναι πώ γίνεται όλο αυτό σε τελική ανάλυση. Και τέλο, ε, επενδύσεις. Και εδώ πιστεύω έχουμε ένα σημαντικό, μια σημαντική έλλειψη. Οι επενδύσεις πιστεύω δεν ε, επικεντρώνονται επαρκώς στην υλοποίηση των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Κάνουμε διάφορες επενδύσεις που προωθούν την αύξηση του ακαθάριστου χώρου προϊόντος μιας χώρας. Πολύ καλό αυτό. Παρ' όλα αυτά, αυτές οι οικονομικές ε, προόδοι πρέπει να εξυπηρετούν και τους πολίτες μιας χώρας. Να τους βοηθούν με κάποιο τρόπο όλες αυτές, ε, όλα αυτά τα μέσα στήριξη, στήριξη στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, διότι δεν μεταφράζονται όλα αυτόματα σε καλύτερη ζωή για τον πληθυσμό. Να ξεφύγει δηλαδή η Αφρική από την παγίδα στην οποία έπεσε η Λατινική Αμερική. Ε, να υπάρχει δηλαδή μια, μια οικονομική ανάπτυξη χωρίς να αμβλύνονται όλο και περισσότερο οι κοινωνικές ανισότητες. Το μήνυμα λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, ε, πιστεύω είναι ανεπαρκές όσον αφορά αυτή την πτυχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ακολουθεί ο κ. Πάγκα που είναι ο εισηγητής μας για τη δική μας γνωμοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επί της Αφρικανικής Στρατηγικής και παρατήρησα ότι πολλές από τις συστάσεις σας ε, συμφωνούν με τις δικές μας ε, και αναφέρομαι τώρα στην εκθεσή μας η οποία θετήθηκε με μεγάλη πλειοψηφία την περασμένη εβδομάδα οπότε συγχαρητήρια. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας στα όσα ακούσαμε σήμερα το μεσημέρι για αυτό το θέμα, παρατηρώ ότι άκουσα πολλά πράγματα τα οποία υπήρχαν και στην έκθεση που υιοθετήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο. Μιλήστε για ε, λυπή πολιτικό διάλογο. Η έκθεσή μας ακριβώς υπογραμμίζει αυτό το αίτημα ενίσχυσης του πολιτικού διαλόγου μεταξύ των δύο υπήρων. Η έκθεση αυτή υπογραμμίζει επίσης το ότι πρέπει να γίνει κάποια διάσκεψη υψηλού επίπεδου στο πλαίσιο αυτού του πολιτικού διαλόγου που θα προσεγγίσει την Αφρικανική και την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Πολλές από αυτές τις πτυχές είναι για μας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βασικοί άξονες οι οποίοι θα συζητηθούν στα τέλη του μήνα στο Αμπιτζάν. Είναι θεμελιώδη σημεία. Ένα από τα σημεία που υπογραμμίσατε ήταν η οικονομική αυτονομία της Αφρικανικής Ένωσης. Θέμα που περιλαμβάνεται και στη δική μας έκθεση να μπορέσει να βρει η Αφρικανική Ένωση χρηματοδοτήσεις που θα της επιτρέψουν να προχωρήσει και να αποδεσμευτεί σε κάποιο βαθμό από τις ε, εξωτερικές αυτές σχέσεις που αναφέρατε στην ε, παρουσίασή σας προηγουμένως. Αυτά ήθελα να πω. Η εκθέσή μας έχει πολλά κοινά σημεία με την δική σας αποτίμηση της κατάστασης. Και υπογραμμίζει για άλλη μια φορά η εκθέση αυτή όλα αυτά τα σημεία τα οποία αναφέρατε εσείς συμπερασματικά στο τέλο των παρεμβάσεών σα. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω όλου του συναδέλφου να ζητούν το λόγο για το θέμα αυτό. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Ξέρω ότι κοιτάτε τη δική μα αξιολόγηση τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική ε, στην Αφρική. Αλλά προφανώ είστε εμπειρογνώμονε στην Αφρική, οπότε θα έχετε δει και άλλε μελέτε Αναρωτιέμαι, έχετε κάνει κάποια σύγκριση ε, με τις ε, σχέσεις που έχουμε για παράδειγμα με την Κίνα και με άλλες χώρες στην Αφρική γιατί ξέρω ε, που έχουν οι Αφρικανικέ χώρε με την Κίνα ή και με εμά. Ε, Μπορείτε να κάνετε τέτοιε συγκρίσει, γιατί ξέρω ότι έχουν σχέσει με την Κίνα πολλέ Αφρικανικέ χώρε. Έχετε πληροφορίε από τι χώρε αυτέ. Πριν σα δώσω το λόγο για να απαντήσετε τι ερωτήσει, λοιπόν, θα ήθελα να καλέσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω αν ε, θέλουν και αυτοί να μα πούν κάτι για τη μελέτη ή για τη Σύνοδο Κορυφή την επόμενη εβδομάδα. Ξέρω ότι ο κ. ήταν εδώ από νωρί ε, είναι ο για το επόμενο θέμα, αλλά ίσω να θέλει να προσθέσει κάτι και για τη Σύνοδο Κορυφή. Δεν ξέρω ποιο θέλει να μιλήσει πρώτο. Είναι και ο κ. Βαν Μέρμπεκ εδώ, ο οποίο πρόκειται να μα πει κάτι για τη μελέτη. Ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να συγχαρώ τους συντάκτες της μελέτης αυτής, γιατί ήταν δύσκολο το έργο τους. Πραγματικά το να μπορεί να, δεις, να ρίξει κανείς μια ματιά ε, σε αυτό το αχανές πεδίο είναι κάτι που μπορεί να δημιουργήσει δέος. Είναι ένα τεράστιο έργο. Αυτό που εγώ βρίσκω δύσκολο σαν τέτοιο εγχείρημα είναι να ορίσει κανείς μέχρι που πηγαίνουμε. Γιατί είναι πολύ ευρεία η εταιρική σχέση. Το 2014, στο πλαίσιο του οδικού 714 εστιάσαμε σε κάποιες προτεραιότητες σε επίπεδο υπήρων και όχι σε σχέση με το τι γίνεται στο πλαίσιο της Συμφωνίας Κοτώνου για παράδειγμα. Και νομίζω ότι αποτιμά θετικά η μελέτη τα όσα έχουμε κάνει. Ίσως λείπει όμως κάτι τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με κάποια προγράμματα και καλό θα ήταν να υπάρχει μια σύγκριση μεταξύ των παλαιότερων και των νέων μέσων και το τι κάνουν τα κράτη-μέλη που και αυτά έχουν συμβάλει στους στόχους ε, του οδικού χάρτη, αλλά καταλαβαίνω πόσο δύσκολο θα ήταν και κάτι τέτοιο. Ελπίζω να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη να καλύτερα όλες τις πτυχές της συνεργασίας μας με την Αφρική όταν κάνουμε μια ευθυγράμμιση στις εμφωνίες Κοτονού με την κοινή στρατηγική Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής. Ευθυγράμμιση και των μέσων και μηχανισμών που έχουμε. Για μετά την περίοδο, από την περίοδο μετά το 2020 έχουμε διαπραγματευτεί την εντολή μας για το Κοτονού. Σίγουρα την επόμενη εβδομάδα στο Αμπιτζάν θα είναι ευκαιρία να έχουμε την πρώτη συζήτηση με τους Αφρικανούς εταίρους εφ' όλων αυτών των πτυχών. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Σε ό,τι αφορά συστάσεις που έχετε διατυπώσει, έχω κάποια σχόλια. Αλλά ίσως να μην είναι καλό να μπούμε σε τέτοιο επίπεδο λεπτομέρειες τώρα και θα μπορούσαμε να το δούμε αργότερα ενδεχομένω. Ίσως και πιο ανεπίσημα. Ευχαριστώ. Α, συγγνώμη για τη διάσκεψη, επειδή ρωτήσατε κυρία Πρόεδρε, ναι, θα ήταν χρήσιμο η κυρία Πρόεδρος να μας πείτε τι προβλέπετε για την επόμενη εβδομάδα. Έχει υπάρξει μια διακήρυξη, διαπραγματεύσει, θα ήταν θετικό να μας πείτε κάποια πράγματα. Και σήμερα και αύριο ε, είναι η συνάδελφοί μου στην αντί για να διαπραγματευτούν ε, το κείμενο της πολιτικής διακήρυξης ε, και τα άλλα έγγραφα που είναι συζήτηση ακόμη και ίσως θα χρειαστεί μέχρι το τέλος εβδομάδας. Υπάρχουν κάποια επίμαχα ζητήματα. Ελπίζουμε να τα έχουμε όμως ε, επιλύσει πριν τη συνεδρίαση της 26ης. Από την παρελθούσα εμπειρία μας ξέρουμε ότι υπάρχουν κάποια καθόδη ζητήματα που μπορεί να μας ε, καθυστερήσουν και στις επισήμες διακηρύξεις. Όπως ε, η καταπολέμηση του φαινομένου τιμωρησίας, ποινική δικαιοσύνη θα υπάρξει 28 μια πρική συνάντηση για τις 29 και 30. Θα συζητήσουμε σημαντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο εταίρων. Δεν είναι επίμαχο. Αλλά σε τα βασικά και τις λεπτομέρειες δεν έχουμε ακόμη καταλήξει ό,τι αφορά τις συγκεκριμένα σημεία των σχέδιων Τετάρτη ο κύριος Τούς και ο κύριος Γιούνκερ θα συναντήσουν ε, τους ε, ομολόγους τους. Προέδρους. Θα είναι και ο πρόεδρος Αφρικανικής Ένωσης. Και εσείς θα κάνετε μια παρουσίαση. Φαντάζομαι θα συζητήσετε την επόμενη εβδομάδα τους κύριους Γιούνκερ και Τούσκ. Back Ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στους ερευνητές μας. Δεν ξέρω ποιος θα απαντήσει. Θα απαντήσω σε κάποια πράγματα όσον αφορά τις πολιτικές πτυχές, ίσως και μετά θα δώσω το λόγο στους συναδέλφους. Πρώτον, όσον αφορά τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η μελέτη έκανε μια συνολική αξιολόγηση της κοινή εταιρικής σχέσης Αφρικής Ευρωπαϊκής Ένωσης και έπρεπε να γίνουν όλα σε 30 σελίδες. Δεν υπήρχε χώρος και δυνατότητα να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες για τα διάφορα χρηματοπιστωτικά μέσα και τη συμβολή του κάθε κράτους μέλους, αλλά φυσικά αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και θέμα άλλης μελέτης επί του θέματος. Αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε στη μελέτη είναι να επισημάνουμε το γεγονός ότι η ίδια η εταιρική σχέση εξακολουθεί να αποτελεί πολύ σημαντικό πλαίσιο για συνεργασία ε, σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ των δύο υπήρων, αλλά φυσικά είναι πολύ ευρεία. Ε, έγινε πριν από 10 χρόνια ε, σε μια χρονική συγκυρία που η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Αφρικανική Ένωση ήταν πολύ διαφορετικές οργανώσεις και η πραγματικότητα επιτόπου και στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αφρική ήταν πολύ διαφορετικές. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε λοιπόν είναι να προωθήσουμε κάποιες ιδέες για την ανανέωση αυτής της εταιρικής σχέσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπάθησε ήδη να το κάνει με την κοινή ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε το Μάιο και θα μπορούσε να θεωρηθεί ε, ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση υπό την έννοια ότι σε αυτή την κοινή ανακοίνωση υπάρχει μια απόπειρα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης να επικεντρωθούν σε πιο συγκεκριμένες προτεραιότητες που είναι σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επομένως να γίνει λίγο πιο στρατηγική η σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής. Το βασικό πρόβλημα όμω με την κοινή ανακοίνωση είναι ότι είναι 100% ένα αυθεντικό ευρωπαϊκό προϊόν το οποίο δεν έγινε από κοινού με τους Αφρικανούς εταίρους και σίγουρα δεν υπάρχει το αφρικανικό όραμα για το θέμα αυτό. Γι' αυτό και είπαμε λοιπόν στην επόμενη σύνοδο, πέραν των όσων ήδη σχεδιάζονται το πολύ σημαντικό θέμα της νεολαίας, της ε, ε, των νέων κλπ, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επικεντρωθούμε και σε αυτές τις βασικές στρατηγικές προτεραιότητες για το μέλλον και επιπλέον, γιατί όχι, να προσπαθήσουμε να βρούμε και κοινό ε, έδαφος για την ανανέωση της εταιρικής σχέσης και ίσως να έχουμε μια νέα κοινή στρατηγική μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και, Αρχή... Ε, και Αφρικής. Όσον αφορά τις θεσμικές ε, πτυχές, συμφωνώ απόλυτα με τα σχόλια τα οποία έγιναν. Υπάρχει ε, το εξή θέμα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και η Αφρική κάνουν συναντήσει σε διαφορετικά επίπεδα και οι συναντήσει σαν επιτροπή είναι πολύ σημαντικέ για να προωθήσουμε συγκεκριμένε τομεακέ πολιτικέ. Αλλά όπω είπαμε, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να εξασφαλίσουμε δέσμευση στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο από τα κράτη-μέλη. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν οι υπουργοί που εκπροσωπούν τις χώρες μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Αφρική συμμετέχουν πλήρως στην εταιρική ε, σχέση. Αυτό προβλεπόταν αρχικά στην εταιρική σχέση, αλλά αν δούμε τι έχει γίνει μέχρι τώρα, ε, αυτές οι υπουργικές ε, ε, συναντήσεις είναι το στοιχείο που λείπει στην εταιρική σχέση με κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα τη Σύνοδο της Βαλέτας, όπου είχαμε σαφώς μια αντίδραση σε μια προτεραιότητα για, μια, για πολλά κράτη-μέλη και υπήρχε μεγάλη συμμετοχή και τα κράτη-μέλη συμμετείχαν ενεργά στην όλη διαδικασία. Αλλά αυτό έγινε εκτός του θεσμικού πλαισίου της ίδιας εταιρικής σχέσης και τα αποτελέσματα αυτής της συνόδου ε, την χάνουν ε, ε μικτών ε, σχολείων από πλευράς κυρίως Αφρικής. Ε, θεωρήθηκε απλώς κάποιος διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Αφρικής και όχι τίποτα περισσότερο. Και τέλος πρέπει να το προσαρμόσουμε στη νέα διεθνή πραγματικότητα και να λάβουμε υπόψη και τον ακτιβισμό των διαφόρων παραγόντων στην Αφρική, ε, πώς δραστηριοποιούνται. Η Κίνα είναι ο υπαριθμόν ένα ανταγωνιστής και πιθανώς και ένας εταίρος που θα μπορούσαμε να λάβουμε υπόψη. Ε, βεβαίως ε, έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να ξεκινήσει ένας διάλογος με την Κίνα και με την Κίνα και την Αφρική για την Αφρικανική Ήπειρο αλλά τα αποτελέσματα είναι ακόμα πενιχρά. Ε, υπάρχουν ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν την προσέγγιση που αναπτύσσει κάθε πλευρά για την Αφρική και η βασική ιδέα της αιρεσιμότητας που είναι ουσιαστική αρχή για την Ευρώπη, ενώ η Κίνα προτείνει ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο, το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, για τους Αφρικανούς ηγέτες. Όσον αφορά την πτυχή αυτή, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μείνει στις βασικές αξίες και προσεγγίσεις που έχει αναπτύξει ε, μέχρι τούδε, αλλά ταυτόχρονα να έχει και πιο δυναμικό πλαίσιο συνεργασίας, ιδιαίτερα σε κάποιους τομείς ε, τους οποίους αναφέραμε προηγουμένως. Για παράδειγμα, ε, διασύνδεση δικτύων, υποδομές, δημιουργίες θέσεων εργασίας και ούτω Αυτά είναι θέματα για τα οποία πιστεύω ότι ότι ένας τριμερής διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικής και Κίνας θα μπορούσε να αναπτυχθεί περαιτέρω. Θέλετε να προσθέσετε και εσείς κάτι εν συντομία. Παρακαλώ. Να είστε σύντομο αν μπορείτε. Λοιπόν, όσον αφορά τους ε, παγκόσμιους ε, παράγοντες, ας πούμε, φορείς που υπέραζουν τα πράγματα, δεν είναι μόνο η Κίνα, αλλά και οι χώρες του κόλπου. Η Ινδία, και άλλοι. Οπότε πρέπει να θεωρήσουμε ότι οι σχέσει Ευρωπαϊκή Ένωση και Αφρική κινούνται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο. Είτε μα αρέσει είτε όχι. Αλλά έτσι είναι η παγκόσμια κατάσταση. Εκτιμώ ιδιαίτερα που η έκθεση εδώ του Κοινοβουλίου περιλάμβανε πολλές από αυτά, πτυχές από αυτά που αναφέραμε και εμείς. Είναι πολύ θετικό αυτό. Ευχαριστώ. Ναι, πολύ γρήγορα για τις επενδύσεις και τη σχέση με τους στόχου βιώσιμη ανάπτυξη Αυτό που μας εντυπωσιάζει ότι αν δούμε τον ε, οδικό χάρτη 2014-2017, η SDG και το κλίμα είναι ένα κομμάτι των προκλήσεων ε, και η εξέταση των επιπτώσεων αυτών των δύο πτυχών ε, ήταν κάτι σημαντικό. Αυτό που προσπαθούμε είναι να συγκεράσουμε αυτά τα δύο θέματα την ανάπτυξη, γενικότερα το κλιματικό ζήτημα, την πρόσβαση σε βιώσιμη ενέργεια, να τα βάλουμε όλα αυτά μαζί και να τα αξιοποιήσουμε δημιουργώντας έτσι ένα πλαίσιο το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στην Ήπειρο να λαμβάνει υπόψη αυτούς τους τρεις παραγόντες, να τους αξιοποιεί ώστε να φτάσει σε πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη και επιπλέον να ε, δημιουργήσει τα ρυθμιστικά και νομικά πλαίσια και θεσμικά πλαίσια τα οποία θα επιτρέψουν να γίνει σύνδεση μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και βιωσιμότητας αυτής της οικονομικής ανάπτυξης. Απλά για να αναφέρω την ενέργεια, ένα από τα βασικά θέματα όσον αφορά τι κινέζικε επενδύσει στην περιοχή, οι οποίε γίνονται μαζικέ, ε, υπερβαίνουν ε, τι δυτικέ όλες τις δυτικές ε, και της Παγκόσμια Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής ε, Τράπεζα Επενδύσεων των κρατών μελών της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως ανέφερε και η Νικολέτα, η ελκυστικότητα των επενδύσεων αυτών είναι πιθανότατα διαφορετική αν τις δει κανείς από την αφρικανική πλευρά. Τι μπορούμε να κάνουμε, να τις συνδέσουμε με ένα πιο δικτυωμένο πλαίσιο με μια ευρύτερη κατανόηση του ενεργειακού ζητήματος που σχετίζεται με το κλιματικό ζήτημα και με το ζήτημα της ανάπτυξης της Υπήρου. Αυτός ίσως να είναι ο καλύτερος τρόπος, ίσως και ο μόνος τρόπος για να κάνουμε τις δικές μας επενδύσεις πιο ελκυστικές σε σύγκριση με τις κινέζικες ή άλλες τις ινδικές ή των χωρών του κόλπου. Ευχαριστώ. Αυτά σίγουρα θα πρέπει να τα συζητήσουμε περισσότερο αυτό το ευρύτερο πλαίσιο στην Αφρική. Ε, θα μιλήσουμε σε λίγο γι' αυτό. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ που μας παρουσιάσετε αυτή τη μελέτη. Θα τη χρησιμοποιήσουμε. Είναι πολύ σημαντική για το δικό μας έργο και για το έργο του κ. Πάγκα αλλά και για την προετοιμασία της Συνόδου Κορυφής της επόμενης εβδομάδας. Ευχαριστούμε πολύ. Ας πάρουμε δύο λεπτά για να αλλάξουμε ομιλητές και να καλέσουμε τον κύριο Ρίντολφ να έρθει εδώ για το επόμενο σημείο. Ωραία συναδέλφοι, πάμε στο σημείο 7. Αφορά και αυτό την Αφρική. Αφορά τα περιθώρια ε, επένδυσης ε, μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Βιώσιμης Ανάπτυξης. Πέρυσι εργαστήκαμε εντατικά ώστε να δημιουργήσουμε το νέο αυτό ταμείο, το EFSD, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Βιώσιμης Ανάπτυξης, με σκοπό επενδύσεις ε, στην Αφρική και σε άλλες χώρες ε, γειτονικές. Ειδικότερα σε χώρες ε, όπου άλλες εμπορικές επενδύσεις δεν πάνε λόγω της υψηλής επικινδυνότητας. Ε, και επειδή αυτές οι χώρες είναι τόσο εύθραυστες, ξέρετε είναι πολύ σημαντικό να γίνουν επενδύσεις και εκεί. Χαίρομαι πολύ που έχουμε εδώ τον Ρομπέρτο Ριντόλφ, θα μας μιλήσει για το EFSD, είναι ένας από τους αρχιτέκτονες του Ταμείου ε, αυτές τις ιδέες ότι πρέπει να γίνουν περισσότερες επενδύσεις. Ακριβώς πριν έρθει ο Ρομπέρτο μας έκανε μια παρουσίαση η UNICEF για τις δημογραφικές προκλήσεις στην Αφρική. Ε, μας είπαν ότι μέχρι το τέλος του αιώνα περισσότερα από τα μισά ε, παιδιά θα γεννιούνται στην Αφρική. Ένα στα 13 στην Ιγυρία και μιλήσαμε για τις υπηρεσίες προς αυτά τα παιδιά αλλά και για το θέμα τη ε, συνόδου τη επόμενη εβδομάδα. Πώ θα παρέχουμε θέσει εργασία και ευημερία στην Αφρική, που είναι η γειτονική μα ήπειρο. Ε, πολύ σημαντική συζήτηση. Και αναμένουμε τη συνόδο και έχουμε τώρα και ένα προσκεκλημένο με μεγάλη εμπειρία από τον ε, ιδιωτικό τομέα, τον κύριο Μάικ Λάντα, Γενικό Διευθυντή τη CTI Global. ήρθε εδώ για να μας πει κάποια πράγματα από την εμπειρία του ως επενδυτή στην Αφρική. Θα σας ακούσουμε σε λίγο. Πρώτα απ' όλα δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Ρίντολφ. Ρομπερτ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Πρώτα απ' όλα ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που συνέβαλε πνευματικά για να γίνει σήμερα αυτό που είναι το επενδυτικό σχέδιο. Το εξωτερικό επενδυτικό σχέδιο σχετίζεται στενά με αυτό που είπατε πριν λίγα λεπτά. Είναι αλληλένδετο με την αναπτυξιακή πολιτική της Ένωσης. Από εμπειρίας γνωρίζω ότι όταν λέμε ότι ο πολιτικός διάλογος δεν λειτουργεί πολύ καλά, Γνωρίζω ότι υπάρχουν και χώρες όπου λειτουργεί και όπου δημιουργείται, σχηματίζεται πρόοδος. Όταν μιλάμε για επενδύσεις, για επενδυτικό κλίμα, για γραφειοκρατία, για διαφθορά και από την άλλη για νομοθεσία ε, που επιτρέπει τις επενδύσεις ε, όλα αυτά είναι ο πυλώνας 3 όπως ξέρετε και μετά ο πυλώνας 1 για τον οποίο συζητήσαμε σήμερα τα πέντε αυτά παράθυρα είναι η οργάνωση αυτών των επενδύσεων. Ε, σε ποιους τομείς, ε, ε, βάσει ποιων συγκεκριμένων προσεγγίσεων θέλουμε να λάβουν χώρα αυτές οι επενδύσεις. Είμαι εδώ λοιπόν σήμερα και σας ευχαριστώ για την γρήγορη διαδικασία για να σας πω ότι είμαστε υπό συνεχή πίεση. Αισθάνομαι κάπως σαν πατέρας του EIP που τώρα είναι σαν ε, ε, παιδί που έχουμε υιοθετήσει και προσπαθούμε να το κάνουμε να προοδεύσει. Όσον αφορά τα δημογραφικά στοιχεία, Λίντα, θα μπορούσε κανείς να θεωρήσει το δημογραφικό θέμα ως θετική πτυχή. Θα υπάρξω πολύ τολμηρό σήμερα το απόγευμα στα όσα θα πω. Οι σημερινές οικονομικές θεωρίες που διδάσκονται στις οικονομικές σχολές αναφέρονται σε κρίσιμη μάζα καταναλωτών για τις, αγοράς, για τις αγορές. Γιατί λοιπόν να μην θεωρήσουμε αυτό το δημογραφικό θέμα θετικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα δημιουργήσουν οικονομική ανάπτυξη. Η δυσκολία είναι η ανάπτυξη αυτή να καταστεί βιώσιμη. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι κατά μέσο όρο θα έχουν περισσότερες ικανότητες και μεγαλύτερη μόρφωση από ό,τι ήμασταν εμείς πριν από 50 χρόνια. Υπάρχει λοιπόν περίπτωση να οδηγηθούμε σε μια καλή κατάσταση, ειδικότερα αν εργαστούμε αποτελεσματικά με στην επόμενη 20 ετία, διότι το 2050 είναι το κρίσιμο έτος όπου θα πρέπει να βρούμε ε, έχουμε δημιουργήσει σχεδόν ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Να σας δείξω σημερινή κατάσταση. 28 Σεπτεμβρίου συζητήσαμε στο Στρατηγικό Συμβούλιο ε, ήταν οι τρεις συζητητές και η Λίντα, ήσασταν και εσείς εκεί. Ε, συζητήσαμε ε, τα Windows αυτά τα παράθυρα, τα οποία εγκρίθηκαν στο σύνολό τους και τέθηκαν και κάποια θέματα που αφορούσαν το, το, το, κανονισμό που θα ακολουθήσουμε. Η γραφειοκρατία πάντα είναι ένα πρόβλημα. 7 Νοεμβρίου Είχαμε τα ε, Συμβούλια εφαρμογή στα Operational Boards και 24 Νοεμβρίου ελπίζουμε να ανακοινώσουμε αυτά τα παράθυρα στη Σύνοδο Κορυφή Εταιρική Σχέσης, διότι ε, μεθαύριο την Πέμπτη η Επιτροπή θα υιοθετήσει αυτά τα παράθυρα, αυτή την απόφαση. Ελπίζουμε λοιπόν να πάνε όλα καλά. 29 Νοεμβρίου θα κάνουμε την ανακοίνωση στη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Αφρικής ε, και θα έχουμε εκπονήσει έναν οδηγό, ένα μικρό εγχειρίδιο αυτή τη στιγμή εκπονείται ώστε να δώσουμε οδηγίες για το πώς θα γίνει το EIP. Έχουμε πολλές ερωτήσεις και δεν έχουν απαντηθεί ακόμα όλες, ούτε υπάρχουν όλες οι λεπτομέρειες, αλλά έχουμε αρκετές πληροφορίες σήμερα για να μπορέσουμε να εξηγήσουμε πώς θα λειτουργήσει το πράγμα. Και αυτό ήθελα να σας εξηγήσω και εσά σήμερα, ώστε να γίνετε πρέσβεις και πρέσβυρες ε, της EIP ε, στους ιδιώτες επενδυτές. Στις 12 Δεκεμβρίου θα παρουσιάσουμε ένα, δύο-τρία παράθυρα που είναι πολύ σημαντικά για μας, η κλιματική αλλαγή και οι, ανα, οι πηγές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ε, το παραθυρό των βιώσιμων πόλεων και η γεωργία και η ευφυής γεωργία. Τέλη Ιανουαρίου μετά θα ζητήσουμε να υποβληθούν ε, το Δεκέμβριο οι προτάσεις. Σε ποιον στα ε, επιλέξιμα, στους επιλέξιμους οργανισμούς. Ποιοι είναι αυτοί. Είναι αναπτυξιακές τράπεζες χονδρικά, ευρωπαϊκές, ε, πολυμερείς EBRD, EAB, Δημερός ε, και FW, Jean Francais, FMO, 15 άλλες και να σας πω ήδη τώρα ότι ήδη από το Δεκέμβριο θα οθήσουμε ε, τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν τους δικούς τους αναπτυξιακούς οργανισμούς. Έχουμε πολύ λίγους, είχαμε 10 ή 12 στα 28 χώρες, θέλουμε να υπάρχουν πολύ περισσότεροι και θέλουμε λοιπόν να καλέσουμε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσουν τμήματα ε, στα δικά τους ε, Υπουργεία για αυτές τις εργασίες, γιατί χρειαζόμαστε πολλούς περισσότερους συμμετέχοντες και φυσικά θα δούμε και τις αναπτυξιακές τράπεζες περιφερειακά στην Νότια, Δυτική, Ανατολική Αφρική. Πρέπει να τους δώσουμε διαπιστεύσεις, να περάσουν μια αξιολόγηση 7 πυλώνων και τα λοιπά, ώστε να γίνουν επιλέξιμες. Αλλά αυτά ε, οι επιλέξιμοι οργανισμοί θα παρουσιάσουν στη συνέχεια προτάσεις. Τι είδους προτάσεις. Ε, οι προτάσεις αυτές θα είναι χρηματοοικονομικά προϊόντα, χρηματοπιστωτικά προϊόντα όπου θα προσφέρουν μέρη των εγγυήσεων σε επιχειρηματίες, σε ιδιώτες επενδυτές, ώστε αυτοί να επενδύσουν στη γεωργία, στην ενέργεια, στην αστική ανάπτυξη κτλ. Έτσι θα λειτουργήσουν τα πράγματα. Με πολλούς και διάφορους λοιπόν συμμετέχοντες στην ανάπτυξη αυτών των χρηματοπιστωτικών προϊόντων, εμείς ως Επιτροπή και όλοι μας θα έχουμε μια επιλογή να επιλέξουμε ότι καλύτερο μπορούμε βάσει των αποτελεσμάτων, δημιουργίας θέσεων εργασίας για παράδειγμα ή επίτευξη των στόχων της κλιματικής αλλαγής, να επιλέξουμε ό,τι καλύτερο απόψη μόχλευσης και ό,τι καλύτερο φυσικά και από άποψη ε, γεωγραφίας Δηλαδή όχι πράγματα που θα απευθύνονται μόνο σε εύκολες χώρες αλλά και πράγματα που θα απευθύνονται σε δύσκολες χώρες γιατί αυτή είναι η εντολή μας ε, για να δημιουργήσουμε αυτή την προσθετικότητα. Αν θεωρήσουμε λοιπόν θα έχουμε λάβει την πρόταση μέχρι τέλη Ιανουαρίου στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις προτάσεις θα θυμάστε την συζήτηση με την EIB, ε αυτή συζήτησα με τους εμπρογνώμενους που εξέτασαν τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές ε, πτυχές. Κινητοποιήθηκαν όλες ε, οι υπηρεσίες της Κομισιόν για να δουν τα κοινωνικά, περιβαλλοντικά και τα πολιτικά θέματα. Θα τα αξιολογήσουμε όλα αυτά. Θα πάμε στο, ε, συμβούλιο, στο λειτουργικό συμβούλιο του Operational Board θα καταθέσουμε μια πρόταση προς έγκριση και θα υπογράψουμε τις συμβάσεις Απρίλιο-Μάιο και αφού υπογραφούν τότε οι συμβάσεις εκείνη τη στιγμή τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εφόσον έχουν ήδη δημιουργήσει Κάποιε επαφέ και τι έχουμε καλέσει να συζητήσουν με ιδιωτικέ επιχειρήσεις. Οπότε το που θα πάνε οι αυτές λοιπόν ε, και πώς ε, θα πρέπει να γίνει αρκετά γρήγορα για να ακολουθήσουν οι πραγματικές επενδύσεις. Και εκεί θα συστήσουμε ένα σύστημα παρακολούθησης που θα επαληθεύει ότι όντως δημιουργούνται βιώσιμες θέσεις εργασίας και θέλουμε να εφαρμοστεί και αυτή η σου επιμέλεια που και εσείς αναφέρετε στον κανονισμό. Να σε εξηγήσω τους πέντε τομείς, τα τέσσερα, τους πέντε τομείς, τα πέντε παράθυρα, τα επενδυτικά παράθυρα, που εγκρίθηκαν με ενθουσιασμό από το Στρατηγικό Συμβούλιο Συνολικής Στρατηγικής. Ε, και το Operational Board ε, έδωσε πολύ καλά σχόλια, πολύ καλή εκτίμηση. Στα πέντε αυτά παράθυρα υπάρχει ένα πράγμα που ονομάζεται μεγάλη εγγύηση κατά του κινδύνου τοπικού νομίσματος. Θα επενδύει κανείς σε ευρώ και, αυτά, και λαμβάνει κανείς τοπικό νόμισμα, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος αποτίμησης. Οπότε όλοι οι επενδυτές ε, αναζητούν κάποια εγγύηση που θα εξισορροπήσει τον κίνδυνο αυτόν. Δεν είναι κάτι εύκολο, είναι κάτι πολύ ακριβό, πολύ περίπλοκο. Γι' αυτό τον λόγο αναζητάμε μια πρόταση που τελικά θα καλύψει όλα τα παράθυρα. Αηφόρος, ενέργεια και συνδεσιμότητα και χρηματοδότηση MSME είναι τα δύο παράθυρα που είναι πιο έτοιμα από ό,τι ακούμε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Θα έχουμε ήδη κάποιες προτάσεις, ε, υπάρχουν ήδη κάποιες προτάσεις σε αυτούς τους δύο τομείς, διότι έχει γίνει ήδη η απαραίτητη δουλειά. Ένα παράδειγμα στον τομέα της, της βιώσιμης ενέργειας είναι η αντικατάσταση της εγγύησης του παραλήπτη. Όταν υπογράφει κανείς μια συμφωνία με μια χώρα Χ, αυτή δεσμεύεται να αγοράσει το ηλεκτρικό ρεύμα, για παράδειγμα με 9 σεντζαλά κιλοβατόρα για 25 χρόνια. Αυτή η εγγύηση μερικές φορές δεν είναι επαρκώς ε, δυνατή και οι επενδυτές ε, που μπορούν να βρουν πολύ φθηνά χρήματα διστάζουν να κάνουν την επένδυση διότι η εγγύηση που προσφέρεται για αυτή την 25 ετία δεν είναι αρκετά ε, βαρύ. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε αυτό το εμπόδιο και να χρησιμοποιήσουμε ε, να εξισορροπήσουμε και το δημοσιοχρέος που δημιουργείται μέσω αυτή τη εγγύηση, παρέχοντα εμεί μια εγγύηση πιο αποτελεσματική. Και η MSME είναι ένα τομέα όπου έχουμε πολλέ προτάσει, ε, ειδικότερα μέσω των EDFI και στις βιώσιμες πόλεις υπάρχουν δύο-τρεις τομείς, η βιώσιμη γεωργία, η ε, αγρότες επιχειρηματίες και οι αγροδιατροφικές επιχειρήσεις είναι σημαντικός ε, τομέας γιατί δημιουργεί περισσότερες θέσεις αναλογικά και μετά το ψηφιακά. Τα ψηφιακά όπως εξήγησα και την περασμένη φορά είναι ένας τομέας όπου κανονικά υπάρχει αγορά για να υπάρξουν επενδύσεις εκεί κοιτάμε την πλατφόρμα για τις μικροπιστώσεις, για τις ψηφιακές υπηρεσίες και μετά οι λύσεις ηλεκτρονικής ε, ε, διακυβέρνησης. Ας τα δούμε στα γρήγορα. Ε, παραγωγή βιώσιμη ενέργεια και προβιώσιμη ενέργεια. Δεν θέλω να μπω σε υπερβολικά πολλέ λεπτομέρειε. Τα βλέπετε όλα εδώ. Πιστεύω με τρόπο αρκετά κατανοητό εδώ έχουμε και δράσει για την ενεργειακή απόδοση, ειδικότερα όσον αφορά τι πόλεις που λαμβάνουν την ενέργεια. Διότι δεν μπορεί να εξοικονομήσει κανεί ενέργεια αν δεν λαμβάνει ενέργεια. Η εγγύηση είναι δομημένη έτσι ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο κίνδυνος, ο πραγματικός και ο ε, αντιληπτός ε, συμπεριλαμβανομένων και των θεσμικών επενδυτών όπως τα συνταξιδοτικά ταμεία. Για να κινητοποιηθούν αυτά πρέπει να δημιουργηθεί ε, κάποια βάση, βάσει των χρημάτων της δικής μας ε, εγγύησης. Ε, πάνω από αυτό δημιουργείται το επόμενο επίπεδο επένδυσης που είναι οι, οι αναπτυξιακές τράπεζες και μετά στο τρίτο επίπεδο έχουμε τα διάφορα συνταξιδοτικά ταμεία με διάφορους κινδύνους χαμηλού κινδύνου, τα μεγάλα χρήματα από σύνταξη οδοτικά ταμεία, μέσος κίνδυνος από τους αναπτυξιακούς επενδυτές και μεγάλος κίνδυνος αυτός που διατρέχουμε εμείς. Ε, εκεί λοιπόν τα 100 μας δισεκατομμύρια μπορεί να γίνουν 2 δισεκατομμύρια επένδυσης. Υπάρχει ένα σύστημα που ονομάζεται Cascade Funding που χρησιμοποιεί διάφορα επίπεδα κινδύνου και που μπορεί να εφαρμοστεί και στα πέντε παράθυρα. Πάμε στο επόμενο, εμείς. Εδώ έχουμε τεράστιες δυνατότητες. Ε, για πολύ ευαίσθητες ε, ε, καταστάσεις. Μιλάμε εδώ για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Σε αυτό το τομέα λέμε συχνά στους συναδέλφους των Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων ότι ξέρετε εδώ μπορεί να χρειαστούν άλλες οργανώσεις. Μπορεί να χρειαστούμε την ΑΕΦΣΥ από την Παγκοσμία Τράπεζα για παράδειγμα. Μπορεί να χρειαστούμε την IFAD, δεν ξέρω αν γνωρίζετε την IFAD, το Διεθνές Ταμείο Γεωργίας και Ανάπτυξης για τους ε, μικρούς γεωργούς που με έδρα στη Ρώμη. Αυτοί έχουν την εντολή. Πρέπει να δεχτεί κανείς λοιπόν ότι όταν περνάμε εδώ στη χρηματοδότηση μικρών, πολύ μικρών, μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, υπάρχει άλλη επικινδυνότητα. Ε, έχουμε εδώ μια ενδιαφέρουσα συνεργασία με έναν οργανισμό που ονομάζεται Cordis. Προωθούμε την αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και μη εμπορικών ε, ΜΚΟ που εργάζονται σε πολύ δύσκολε περιοχέ, όπω α στη Σομαλία. Δεν μπορεί φυσικά να έχει κανεί την ίδια δομή ε, για τι μικρομεσαίε επιχειρήσει στο Ναϊρόμπι και στη Σομαλία ή στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Πρέπει να ε, αντιληφθεί κανεί ότι υπάρχουν διαφορετικά κίνητρα, διαφορετικέ απαιτήσει προστασία. Ε, και το μέσο ωστόσο αυτό είναι πολλά υποσχόμενο, διότι όπω είπα είναι αναπτυσσόμενο και όπω είπα η δημιουργία θέσεων εργασία είναι πολύ μεγάλη σε αυτο τον τομέα. Ας πάμε στη βιώσιμη γεωργία επιχειρηματίες στις αγροτικές περιοχές και οι σχετικές επιχειρήσεις. Εδώ θέλουμε να υπάρξει μεταρρύθμιση, μετασχηματισμός. Και είναι ένας τομέας εδώ που πραγματικά μπορεί να υπάρξει τεράστιος μετασχηματισμός, τεράστιες αλλαγές αν έχουμε, ας χάρη, μετά την εσοδεία, ε, την επεξεργασία, που καταλήγουν να είναι πολλά τα απορρίμματα και τα απόβλητα, αποθήκευση. Όλα αυτά θα αυξήσουν την προσθέμενη αξία και θα παραμείνει καλή τιμή για δύσκολους καιρούς. Σχεδόν έχω ολοκληρώσει γιατί θέλω και εγώ να έχουμε μια συζήτηση. Ξέρω πώς λειτουργεί εδώ το σύστημα. Έχουμε πει στο Ταμείο που παρέχει ένα τμήμα, ένα κομμάτι της εγγύησης. Πολύ συχνά οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί ζητούν να υπάρξει ένα μείγμα πόρων. Έχουμε λοιπόν το λεγόμενο blending και προέρχονται πόροι από άλλα κονδύλια και φυσικά υπάρχουν και τεχνική βοήθεια και έχουν ολοκληρωθεί μελέτη σκοπιμότητας για τις επενδύσεις. Βιώσιμες πόλεις πολύ σημαντικό επενδυτικό σκέλος. Έχουν ήδη έρθει σε επαφή μαζί μας κάποιες οργανώσεις. Bloomberg. Είχαμε συναντήσεις και συζητήσεις μεταξύ Μπερτή και Bloomberg, γιατί έχουν πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, ε, ιδέες, συγγνώμη. Θέλω να σας πω και σας ζητώ την υποστήριξή σας για ένα παιδαγωγικό ρόλο για τους χρηματοπιστικού οργανισμούς να φύγουμε από τον τεζαβί και τα απλά πράγματα. Εγγύηση για τις επενδύσει και τίποτα παραπάνω. Να περάσουμε σε κάτι πιο επιτιθευμένο, πιο πολλά υποσχόμενο. Καλό είναι να μην έχουμε μόνο τους συνήθει υπόπτους, αλλά και άλλους παράγοντες. Για να δείξουμε ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι διάρθρωσης αυτών των ε, προϊόντων και προγραμμάτων εγγύσεων για να αναπτυχθούν νέα προγράμματα από νέους εταίρους. Στις βιώσιμες φορές πόλεις εδώ βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά περιθώρια επενδύσεων για τη δημιουργία περιφερειακών στοιχείων. Και το τελευταίο είναι ψηφιακό επίπεδο, ψηφιακό τομέα για την ανάπτυξη. Digital for development. Υπάρχει έντονο ψηφιακό χάσμα. Αν έχουμε λοιπόν διαδικτυακές λύσεις με τις σχετικές πλατφόρμες μπορούμε να έχουμε και ένα καταλητικό ρόλο για περισσότερες επενδύσεις. Η τελευταία φράση που είναι η ίδια πάντα σε όλα τα επενδυτικά σκέλη, λέμε ότι η εγγύηση θα είναι διαρθρωμένη κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μειώνει τη χρηματοδότηση επενδυτικού κινδύνου και να δημιουργεί τις συνθήκες που θα οδηγήσουν σε περισσότερες ψηφιακές υποδομές. Εδώ θα σταματήσω με την άδειά σα, κύριε Πρόεδρε, ώστε να ακούσω τι ερωτήσει, τι οποίε θα προσπαθήσω να απαντήσω. Ευχαριστώ. members, going... Πριν δώσω το λόγο στα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής μας, θέλω να δώσω τον λόγο στον κύριο Μίχαλ Αντάου, που είναι μέσα στο CTI και έχει νομίζω δουλέψει για πολλά χρόνια και θα μπορούσε να μας πει ακριβώς για την Αφρική και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εκεί, αν θεωρεί ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά, μπορεί να γίνουν και άλλα. Τέλο πάντων, να μα ε, μεταφέρει τι δικέ σα εμπειρίε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να σα συγχαρώ εσά, ως Ευρωπαίους γιατί έχετε ένα πραγματικά ε, μακρόπνο σχέδιο αναπτύξει σε σχέση και με τα άλλα που έχουν αναπτύξει διάφορες χώρες. Ε, αλλά ε, το ότι δεν εστιάζεται στη μετανάστευση. Σας δίνει βέβαια την εστίαση, γιατί βλέπετε ότι το πρόβλημα είναι ολιστικό και θα πρέπει να βρεθεί μια ολιστική λύση για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας στις αφρικανικές χώρες, στις χώρες ε, καταγωγής. Ε, όχι για την καταπολέμηση του φαινομένου της μετανάστευσης, αλλά και της ριζοσπαστικοποίησης. Ε, σας ε, συγχαίρω λοιπόν και ακόμη και η παρουσίαση που ακούσαμε από τον Γενικό Διευθυντή. Οι σιλό υπάρχουν, στεγανά υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι τυπικό, χαρακτηριστικό, όπως κάνουν οι τράπεζες επενδύσεις που κοιτάνε αυτά τα σιλό, αυτά τα στεγανά, αλλά νομίζω ότι πραγματικά έχετε πάρει τα ενία και δημιουργείται μια ολιστική προσέγγιση και αυτό χρειάζεται. Η δική μου εταιρεία ήταν από αυτές που δημιούργησαν την πρώτη κινητή τράπεζα, το MCNT, το 2007 στην Αφρική. Το 2012 ξεκίνησαμε ένα πρόγραμμα που λέγεται The Joseph Initiative, 10.000 ε, ε, μικρούς ε, κτηματίες, μειώσαμε τις απώλειες και τις μηδενίσαμε κιόλας και γενικά έχουμε μεγάλη εμπειρία από τη βάση. Εργαζόμαστε στη βάση της πυραμίδας. Κάτι που ακούστηκε και η θεσμερική συζήτηση, δεν ξέρω αν το είπε η UNICEF ή αν ο ε, συνάδελφος ε, δικός σας ο Ευρωβουλευτής πριν, πράγματι υπάρχουν περιορισμένοι πόροι και θα πρέπει να υπάρξει μόχλευση, άρα μεγιστοποίηση των λίγων διαθέσιμων κονδυλίων και η όλη έννοια πίσω από το EFSD ακριβώς αυτή είναι. Δηλαδή παίρνουμε λίγα χρήματα, μόχλευση, ε, εκμετάλλευση δηλαδή των πηγών από την ιδιωτική βιομηχανία. Και η ίδια είναι και η δική μας προοπτική. Πώς δηλαδή μπορούμε να μοχλεύσουμε από μικρά ε, κονδύλια για να ενισχύσουμε την ε, επίπτωση. Και το δεύτερο είναι τα δεδομένα. Πώς μετράμε τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Πώς γνωρίζουμε αν είναι επιτυχημένη η προσέγγιση μας για την επίτευξη των στόχων. Η CTI έχει αναπτύξει, θα έλεγα, ένα μοναδικό project Πάνω από δεκαετή ήταν η εμπειρία, η δεκαετή ήταν η εμπειρία που χρειάστηκε. Και εστιάζουμε κυρίως στους ε, πολίτες, στις τοπικές κοινωνίες και όχι απαραίτητα στις κυβερνήσεις ή τη στήριξη αυτών και άλλων μεγάλων οργανισμών. Γιατί πιστεύουμε ότι τη δύναμη πρώτα απ' όλα πρέπει να τη βρούμε στους πολίτες, στη βάση. Άρα η ισχύ, όπω και στον ηλεκτρισμό είναι το σημαντικό, και τα δεδομένα το δεύτερο σημαντικό. Χωρί ισχύ δεν γίνεται τίποτα και χωρί δεδομένα επίση δεν γίνεται τίποτα. Έτσι έχουμε αναπτύξει ένα επιτευμένο πρόγραμμα τη συλλογή δηλαδή πολύ σοβαρών δεδομένων. Στην Ουγκάντα και στο Μαλάουι δραστηριοποιούμαστε αυτή τη στιγμή και έχουμε εστιάσει διάφορα πιλωτικά προγράμματα. Χίλιες οικογένειες, 5.000-6.000 άνθρωποι δειγματοληπτικά και εστιάζουμε στο σπίτι και στο χωριό, ληστικά, στο σπίτι, για την ε, ηλιακή ενέργεια, ε, πόσιμο νερό, καθαρό νερό, δηλαδή ό,τι έχει να κάνει με τη, τα υγειονομικές συνθήκες, άνθρωποι που δεν έχουν πόσιμο νερό, που δεν έχουν πρόσβαση στην ενέργεια. Θέλουμε να λύσουμε αυτά τα προβλήματα. Τους δίνουμε και ένα ελεύθερο smartphone, ένα δωρεάν smartphone επίσης. Αν υπάρχει βέβαια ένα μικρό ε, δίκτυο θα τους δώσουμε επίσης ε, και ασύρματη σύνδεση και θα εστιάσουμε σε τρεις βασικούς τομείς. Το συζητήσατε και εσύ, UNICEF ε, και άλλοι το Ένα telemedia center, ό,τι δεδομένα έχουμε συλλέξει, είτε πρόκειται για εγγραμματισμό, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν 30% αναλφάβητοι, ή αυτοί που δεν έχουν ελεγχθεί για AIDS δεν είναι βέβαια έτοιμα όλα αυτά τα στοιχεία, δεν ήταν γρήγορη αρκετή ομάδα για να έχουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Τέλο πάντων, κάποια τέτοια δεδομένα θα συλλέγουμε είτε για τον τομέα τη γενική ε, περίθαλψη, είτε τη παιδεία, είτε τη γεωργία, τη επαγγελματική κατάρτιση. Θα υπάρχει μια σχετική μονάδα και μέσω του smartphone θα υπάρχει δυνατότητα άμεσης πρόσβασης το telehelp μετά, telemedicine, τηλεγιατρική. Τεχνολογικές εξελίξεις είναι τέτοιες σήμερα που μπορούμε στις πιλωτικές αυτές περιοχές να βοηθήσουμε να υπάρχουν ηλεκτρονικά αρχεία και η σωστή ιατρική εξέταση. Να υπάρχει πρόσβαση μέσω του smartphone επίσης. Και πολλά διαγνωστικά τεστ μπορούν να γίνουν απομακρυσμένα. Μέσω του υπολογιστή μη επεμβατικά ή με την ελάχιστη δυνατή ε, παρέμβαση. Ένα νέο μοντέλο δηλαδή παροχής υπηρεσιών υγείας και αυτό ως επιχείρηση. Είμαστε πραγματικά ενθουσιώδεις. Όλοι λένε για τον ιδιωτικό τομέα ότι είμαστε ανέστητοι και το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το κέρδος. Αν δείτε όμως ε, ε, τι γίνεται σε εμά. Δεν είμαστε στο Λονδίνο και στη Νέα Υόρκη προσπαθούμε να κερδίσουμε χρήματα, αλλά προσπαθούμε να βρούμε ολοκληρωμένε λύσει. Τώρα, επειδή δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά θα έρθω στο τρίτο σημείο, το είπε και ο Ρομπέρτο πριν. Γεωργία. Εφής Γεωργία, μας ενδιαφέρει και αυτό. Με αυτά τα δεδομένα που θα συλλέξουμε θα ξέρουμε τι γη έχουν, πόσοι γη καλλιεργούν οι άνθρωποι εκεί, τα ζυζανιοκτώνα, τα φυτοφάρμακα, τους εμπορικούς σπόρους ε, που χρησιμοποιούν. Και έτσι θα μπορούμε να είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί για να τους παρέχουμε τους σωστούς σπόρους και τα σωστά λοιπάσματα. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τους εκπαιδεύσουμε τους στέλνουμε στο κέντρο της κοινότητας για να παρακολουθήσουν το σχετικό παιδευτικό γεωργικό πρόγραμμα. Και στο smartphone θα τους ε, θυμόμίζουμε πότε πρέπει να ποτίσουν, ε, πότε πρέπει να κάνουν άλλα που μπορεί για μας να είναι αυτονόητα. Τέλος πάντων, ε, ο στόχος είναι να παρέχουμε εκτεταμένες υπηρεσίες και παρά τι πολλέ προσπάθειε που έχουν γίνει μέχρι τώρα ο κόσμο δεν έχει εκπαιδευτεί επαρκώ. εμεί θέλουμε να εκπαιδεύσουμε του αγρότες και για καλύτερη εισοδεία. Και αν ξέρουμε τι καλλιεργείται, θα μπορούμε να προδικάζουμε, να προβλέπουμε τι ε, θέλει η αγορά και να ενημερώνουμε σχετικά του αγρότε. Άρα θα μπορούσαν να διπλασιάσουν και να τριπλασιάσουν το εισόδημά του. Μπορεί να κερδίσουν χίλια και να χάνουν 300-400 και θέλουμε να τους βοηθήσουμε από τα 1.000 να φτάσουν στα 1.500 και στα 2.000 να μειώσουν αυτές τις απώλειες λόγω εσοδείας και αυτό σε εθνικό επίπεδο. Το μεταναστευτικό πρόγραμμα. Επίσης ε, δημιουργεί θέσεις εργασίας και στο δικό μας πρόγραμμα θέλουμε να δημιουργήσουμε 6-7 ε, θέσεις εργασίας σε κάθε συγκεκριμένο μέρος, στο συγκεκριμένη τοποθεσία και σε σχέση με τη Γεωργία. Και σε πλήρη συνεργασία με τις κυβερνήσεις εργαζόμαστε σε σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα γίνεται αυτό. Θέλουμε να είμαστε αηφόροι και βιώσιμοι. Δεν είναι ο στόχος μας ε, να πάρουμε την επιδότηση, να την ε, δαπανίσουμε και να φύγουμε. Θέλουμε να μείνουμε πολλά χρόνια. Θέλουμε αηφορία μακροχρόνια. Το CTI λοιπόν με τη δική μας εμπειρία, όπως ε, την έχουμε αποκτήσει την τελευταία δεκαετία, έτσι θέλουμε να προχωρήσουμε. Αλλά δεν θα μείνουμε στα πιλωτικά προγράμματα. Μας αρέσει και αυτό βέβαια, αλλά το θέμα είναι να βελτιώσουμε ε, τη βιωσιμότητα ε, του μοντέλου, την κλίμακα του μοντέλου. Έχουμε 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και για να τους πετύχουμε θέλουμε βοήθεια για να πάμε στο επόμενο επίπεδο. Να ε, ανέβουμε κλίμακα, να πάμε σε εθνική, για να μην πω βέβαια και υπερβάλλω, θα είμαι υπερβολικό παναφρικανική κλίμακα. Τέλο πάντων, ε, αυτά είχα να πω και θέλω να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έκανε μια τόσο ευφύ πρόταση. Να κάνω μια ερώτηση απλώς για τον τρόπο. Μα είπατε ότι είναι πιλωτικό πρόγραμμα. Πού δραστηριοποιείστε, σε ποιε χώρες, σε επίπεδο χωριών, πόλεων, για να είναι λίγο σαφέ αυτό. Ξεκινήσαμε σε δύο χώρες, ε, ε, στην Ουγκάντα, σε μια περιοχή που λέγεται Μποίκουε, είχαμε 7 χωριά, 258 οικογένειες και έχουμε συλλέξει και τα στοιχεία για το 98,3%. Έχουμε 150-160 ερωτήσεις. Υπάρχει σύστημα με τον τρόπο που γίνεται. Ο κόσμος με τα χαράς δίνει τις πληροφορίες και οι κυβερνήσεις τώρα που είδανε τα ε, στοιχεία και τις πληροφορίες που συλλέξαμε, μας ρώτησαν πώς μπορούμε να συνεργαστούμε, γιατί ποτέ δεν είχαμε τόσο καλά στοιχεία. Είναι ένας συνδυασμός αξιοπιστίας και μιας προβολής του οράματος ε, που ε, θέλουμε να υλοποιήσουμε αν συνεργαστούν μαζί μας. Και επίσης έχουμε και ένα μικρό χωριό αντσόη στο Μαλάουι που έχει περίπου χίλιες οικογένειες πάνω κάτω. Έτσι είναι λίγο πιο σαφές πώς εργάζεται επί τόπου. Έχω πολλούς ε, συναδέλφους που θέλουν να θέσουν ερωτήσεις στον κύριο Λάντο και στον κύριο Ριντόλφη. Έξι ομιλητές, έχουμε χρόνο, άπλετο, τρία λεπτά ο καθένας το πολύ. Ο Πολ Ρούμπικ είναι ο πρώτος ομιλητής. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι πλέον φτάνουμε σε ένα στάδιο που μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε ότι έγινε καλή διαπραγμάτευση εγκαίρως και είναι και πολύ καλή επιτυχία και από πλευρά τη αναπτυξιακή πολιτική να μπορέσουμε να περάσουμε πραγματικά στον τομέα των επενδύσεων. Για μα είναι πάρα πολύ σαφέ ότι η βασική προτεραιότητα είναι η στόχη τη βιώσιμη ανάπτυξη. Θεωρώ λοιπόν ότι οι καλύτερε επενδυτικέ δραστηριότητε είναι στο στόχο 2, 6 και 7. Ο 2 είναι τα τρόφιμα. Για να ζήσει κανείς χρειάζεται τροφή. Ε, και υπάρχει και ένα πάνελ ε, αξιολόγησης της ε, επιστημονικής ε, ε, τεχνολογίας, το ΣΤΟΑ. Ε, κάναμε μια μελέτη. Το 2030 θα είμαστε περίπου 10 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε αυτό τον πλανήτη. Τι σημαίνει όμως να έχουμε 10 δισεκατομμύρια και υπάρχει αρκετό νερό για να μπορέσουμε να έχουμε όλα αυτά τα γεωργικά προϊόντα που χρειαζόμαστε. Υπάρχει αρκετό νερό για να φτάσει στα νοσοκομεία. Ε, να υπάρχει καθαρό νερό για να μειώσουμε και το κοινωνικό κόστος. Και φυσικά οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο, διότι χωρίς ενέργεια δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη προς τη σωστή κατεύθυνση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ότι κάθε πρόγραμμα χρειάζεται μια συγκεκριμένη αρχιτεκτονική δομή, μηχανική που θα αναπτύξουν το πρόγραμμα, δηλαδή και πρέπει να αναπτυχθεί το καλύτερο πρόγραμμα. Χρειαζόμαστε ένα μοντέλο τριών σταδίων. Πρώτα η αρχιτεκτονική δομή του προγράμματος, δεύτερον να υλοποιηθεί το πρόγραμμα και ε, από εκεί και πέρα να εδραιωθεί αυτό το πρόγραμμα, διότι αυτό το οποίο διδαχθήκαμε μέχρι τούδε είναι ότι πολλά προγράμματα δεν υλοποιούνται γιατί δεν γίνεται κατάλληλη συντήρηση προς τη σωστή κατεύθυνση. Ε, πιστεύετε λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε και τη συντήρηση στο οικονομικό σκέλος. Να έχουμε δηλαδή τρία στάδια. Πρώτο στάδιο ε, δημόσιος διαγωνισμός για την αρχιτεκτονική δομή του προγράμματος, δεύτερον η υλοποίησή του και τρίτον η συντήρηση του προγράμματος. Ε, σε όλους τους τομείς που έχουμε νομίζω ότι θα ήταν καλό να υλοποιηθεί αυτό. Και ένα τελευταίο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε το λεγόμενο πρόγραμμα των Ευρωβουλευτών, ε, ελέγχου, επιστήμονες μαζί με τους ευρωβουλευτές συνεργάζονται για κάποια θέματα. Ο εταίρος μου ήταν η UNESCO ε, και το Πανεπιστήμιο στο Ντέλφτ ε, και μάθαμε πολλά πράγματα για τα προβλήματα στην Αφρική που προκύπτουν από μολυσμένο νερό. Ε, πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα ισοτήμων μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αφρικανικό επίπεδο. Να δούμε την εμπειρία σε επίπεδο μικρών επιχειρήσεων και να το αναβαθμίσουμε από εκεί και πέρα, να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη, να μπορούν να μάθουν ένας από τον άλλον επαγγελματική εκπαίδευση και να έχουμε ε, και γνώσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Νόιζερ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος του εισηγητή, του κυρίου Φραντσούλικα πρέπει να παραμείνει στη Ρουμανία. Δεν μπόρεσε λοιπόν να έρθει εδώ στη συνεδρίαση. Και μου έγραψε ότι ως εισηγητής ε, χαίρεται που ο πρόεδρο τη Επιτροπή ΔΕΒΕ, εσύ δηλαδή Λίντα, η συνάδελφα από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και την Επιτροπή Προπολογισμών ε, συμμετείχαν στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο το Σεπτέμβριο μετά από τη δημοσίευση ε, στην επίσημη εφημερίδα. Ευχαριστούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την κατάλληλη προετοιμασία τη συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου και το γεγονό ότι δόθηκαν οι κατάλληλε πληροφορίε. Το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο έχει συγκληθεί στην ε, συνεδρίαση του Στρατικού Συμβουλίου συζητήθηκε και στον τριμερή διάλογο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό διότι το Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια ανησυχεί διότι υπάρχουν ε, πολλά ε, ειδικά μέσα τα οποία συστήθηκαν με ειδικέ διαδικασίες και διοικητικά συμβούλια, διοικητικούς φορείς, για παράδειγμα η διευκόλυνση για την ε, Τουρκία και τα διάφορα καταπιστεύματα που ε, κάνουν πολύ δύσκολο τον έλεγχο από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ε, τουλάχιστον με καθεστώς ε, παρατηρητή στο Διοικητικό Συμβούλιο μπορούμε εμείς ως μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου να παρακολουθήσουμε τις διάφορες αποφάσεις στη διαδικασία εφαρμογής πιο στενά. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει να συζητήσουμε και όλες αυτές τις αποφάσεις ε, εδώ στην Επιτροπή μας για να διασφαλίσουμε διαφάνεια, λογοδοσία και να είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η διαδικασία θα συνεχίσει να βέβαιει προς τη σωστή κατεύθυνση. Όπως ε, και τα περισσότερα μέλη του Στρατηγικού Συμβουλίου βλέπουμε ε, με χαρά ότι τα πέντε παράθυρα επενδύσεων ακολουθούν τις κατευθυντήρες γραμμές που καθορίστηκαν στις ε, θέσεις του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, οι οποίες παγιώθηκαν από εκεί και πέρα στον τριμερή διάλογο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Αφρική και την γείτονα περιοχή με πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες και πολύ μικρές επιχειρήσεις και αυτό φυσικά ε, είναι πολύ σημαντικό για την επιλογή του πρώτου επενδυτικού παραθύρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την όθηση για νέες επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, αυτό ήταν θέμα συζήτησης στους τριμερείς διαλόγους και ε, το Κοινοβούλιο έδωσε ιδιαίτερη προτεραιότητα σε αυτό και αυτό αντανακλάται στο επενδυτικό παράθυρο 2, την ενέργεια και τη συνδεσιμότητα και στο 3 βιώσιμες πόλεις. Οι επενδύσεις στην επισητιστική ασφάλεια και τη στήριξη προς τους ε, μικρούς γεωργούς και πρόσβαση στη χρηματοδότηση και στις αγορές αποτελούν προτεραιότητα για την Επιτροπή μας εδώ και πάρα πολύ καιρό και καλωσορίζουμε λοιπόν το επενδυτικό παράθυρο 4, ε, γεωργία, για τους ε, μικρούς ε, επιχειρηματίες και τον ε, γεωργικό διατροφικό τομέα. Και επίσης σημειώσαμε στο παρελθόν ότι κίνδυνοι όπως για παράδειγμα η αρπαγή γης θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και να τους αποφύγουμε με κάθε κόστος. Τέλος, το παράθυρο 5 θα πρέπει να βοηθήσει να μειώσουμε το ψηφιακό χάσμα, το οποίο εξακολουθεί να χωρίζει το μεγαλύτερο τμήμα της Αφρικής με τον υπόλοιπο κόσμο ε, για την οικονομία και τα συστήματα πληροφορικής. Ε, στις αφρικανικές χώρες στις οποίες έχει αναπτυχθεί το διαδίκτυο και οι τηλεπικοινωνίες με πιο δυναμικό τρόπο, οι δυνατότητες για βιώσιμη ε, ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς είναι αποδεδειγμένες. Δεν θα πρέπει λοιπόν να επικεντρωθούμε σε προγράμματα στις προ, προηγμένες οικονομίες ε, στην Αφρική, ε, θα πρέπει να κάνουμε τη διαφορά με την αγορά και τις τράπεζες εκεί που δεν θα πήγαιναν πλέον ε, να υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες θεωρούνται πιο επικίνδυνες λόγω του κόστους και εδώ κατάλαβα και αυτό που είπατε όταν αναφερθήκατε ε, σε αυτό τον κλιμακωτό το κίνδυνο Βάδα, στο cascade ε, Νομίζω ότι είναι πολλά υποσχόμενη όλη η διαδικασία. Θα παρακολουθούμε τα προγράμματα τα οποία θα υποστηρίξει το MSD αυτή τη στιγμή και θα δούμε και τι ακριβώς θα γίνει και θα δούμε κατά πόσο τα προγράμματα θα αποτελέσουν πραγματική αξία για τις διάφορες περιοχές και τους ανθρώπους και τις χώρες της Αφρικής, κυρίως τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Επίσης θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε και τον αντίκτυπο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τα πρότυπα διαφάνειας και τα οποία εγγράφονται στον κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά ήταν εκ μέρου ε, του κυρίου Φρουντζούλικα, αλλά αυτή είναι και η θέση τη ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρενς. Ναι, ευχαριστώ. Ο κύριος Ριντόλφη επέμεινε ότι οι επενδύσεις ε, προκύπτουν βάσει εγγυήσεων για τις επενδύσεις και αναφερθήκατε σε έναν από τους κινδύνους που είναι οι διακυμάνσεις στο τοπικό μοντέλο. Θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον στην ε, περιοχή της ε, Δυτικής Αφρικής, ε, στην περιοχή της Δυτικής Αφρικής που κυρίως ενδιαφέρεται για το ευρώ και την ισοτιμία του ευρώ ο, δεν υπάρχει τέτοιος κίνδυνος. Ε, εσείς δηλαδή ουσιαστικά ε, δίνετε προτίμηση σε αυτές τις επενδύσεις, διότι αν πρέπει να εγγυηθούμε για μια επένδυση, αν μπορούμε να έχουμε μηδενικό κίνδυνο, έχετε απεριόριστες δυνατότητες ε, παρέμβασης. Επομένως, τι προσδοκίες έχετε θα αποφύγετε τους πιο σημαντικούς κινδύνους ε, για να επικεντρωθείτε σε περιοχές όπου δεν είναι τόσο σημαντική αυτή η κίνδυνη. Ε, αυτό δεν θα αποτελεί διάκριση υπέρ μιας περιοχής ή μιας χώρας ε, ή μιας κοινότητας επειδή ακριβώς θα παρουσιάζει ψηλότερο κίνδυνο για τις επενδύσεις. Ευχαριστώ κυρία Χόιμπουχ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Λίντα για τον κύριο Ριντόλφη. Όπως ξέρετε αυτό το οποίο ιδιαίτερα με ενδιαφέρει είναι το επενδυτικό ταμείο για την Ήπεθρο, για την ανάπτυξη Πέθρου και ήδη και πριν τις θερινές διακοπές είχα απευθύνει μια γραπτή ερώτηση στην Κομισιόν και εξακολουθώ να περιμένω την απάντηση. Δεν ξέρω μήπως την πάρω τώρα προφορικά από εσάς απευθείας. Και η ερώτησή μου ουσιαστικά είναι ότι από τη μία πλευρά έχουμε το Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα νέο σημαντικό εργαλείο ε, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας ε, και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να στηρίξει τις ε, ευφυείς και καινοτόμες γεωργικές μεθόδους. Εσείς μιλήσατε για, τις, για τη δημογραφική αλλαγή, αλλά πρέπει να την αναφέρεται ως ευκαιρία, αλλά για να είναι ευκαιρία νομίζω ότι θα πρέπει ε, να επενδύσουμε σε αυτό το τομέα, στην Γεωργιακή. Και το ερώτημα που έχω είναι η... αυτό το επενδυτικό σκέλος, οι δυτικές επενδύσεις, συνεταιρισμούς, ε, μικρές ε, γεωργικές εκμεταλλεύσεις μπορεί να είναι πιο αποτελεσματικό και είχαμε και μια συζήτηση, μου είχατε επιβεβαιώσει ότι σε αυτές τις μικρές γεωργικές δομές ε, θα πρέπει να υπάρξουν περισσότερες επενδύσεις, να επιμηκυνθούν οι επενδύσεις. Πώς θα το πετύχετε αυτό. Έχουμε τη νέα συμμαχία για την ασφάλεια που συμμετέχει εκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι διδάγματα έχουμε αντλήσει. Στην έκθεσή μας ασκήσαμε έντονη κριτική σε ό,τι αφορά τη βιομηχανική ε, γεωργία, ότι απειλείται η βιοπικιλότητα, ότι βλάπτονται περισσότερο οι μικροί ε, γεωργοί, δεν χρησιμοποιούν τόσο πολύ αυτές τις δυνατότητες. Έχουμε το land grabbing. Άρα, τι έχουμε διδαχθεί από αυτή τη νέα συμμαχία, από αυτόν τον νέο συνασπισμό, τι μπορούμε να διδαχθούμε για αυτό το σχέδιο εξωτερικών επενδύσεων Πώς μπορούμε να καλύψουμε αυτά τα σφάλματα, πώς ε, θα αποφύγουμε την μάλεψη των σφάλματων αυτών και σε το land grabbing, την αρπαγή των γεών, υπάρχει επιτροπή ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα που παρουσίασε μία μελέτη πριν από κανένα μήνα που λέει ότι μεταξύ άλλων η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, με, τα κριτήρια, με τις επενδύσεις και τις επιδοτήσεις που προσφέρει ουσιαστικά συνεισφέρει στο land grabbing, αυτό που δείχνεται από μελέτες. Σε τέτοιες περιπτώσεις έχει να κάνει και με ιδιωτικούς αλλά και με δημόσιους φορείς. Λένε οι συντάκτες ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός υποβολής καταγγελιών. Πώς θα λειτουργούσε στο Ευρωπαϊκό Επενδυτικό Σχέδιο ένας τέτοιος μηχανισμός θα μπορούσε να συμπεριληφθεί, το συζητείτε καθόλου αυτό. Η Χάιντι αλλά επίση, συνάδελφο που χρειάστηκε να αποχωρήσει νωρίτερα, μου άφησε κάποιε ε, ερωτήσεις τέλος διαφορετικού χαρακτήρα σε ό,τι αφορά τη διαφθορά και τη φοροαποφυγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα διασφαλίσει σε ό,τι αφορά αυτά τα σχέδια του επενδυτικού προγράμματος. Πώς δεν θα γίνει φοροαποφυγή, φοροδιαφυγή, πώς θα αποφευθεί. Υπάρχει ένας μηχανισμός Κάτι όπως και για το land grabbing που προείπα, να μην υπάρξουν καταχρήσεις. Ευχαριστώ. Okay, thank you. Uh, Mr. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σαφάζα. Merci. Ευχαριστώ. Πρώτη αντίδραση πολύ θετική για όλη αυτή την προσέγγιση. Θεωρώ ότι η ουσία του ζητήματος είναι το ερώτημα του πώς δημιουργείται πλούτο σε τοπικό επίπεδο. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Εγώ προέρχομαι από μια πολύ απομακρυσμένη περιοχή, απομονωμένη περιοχή της Αλσατίας και μας λένε οι δρόμοι έκαναν την ανάπτυξη. Όχι. Οι δρόμοι πολλαπλασίασαν τη δημιουργία πλούτου σε τοπικό επίπεδο. Αν δεν υπήρχε ήδη δημιουργία πλούτου, ο δρόμος θα μας χρέωνε περισσότερο και στην Αφρική μετά από 25 ετή ε, εμπειρία το λέω ως ε, πρόεδρος ε, διαφόρων ιδρυμάτων ανάπτυξης έχουμε να κάνουμε με αυτό το πρόβλημα των ατέρμονων στηρίξεων διότι δεν δημιουργούμε επαρκή πλούτο τοπικά. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Πιστεύω λοιπόν ότι πολύ καλά κάνει η Κομισιόν που εξετάζει αυτό το πρόβλημα και προσπαθεί να βρει λύσει. Πώ δηλαδή να δημιουργήσει δραστηριότητε και από αυτέ πλούτο στο τοπικό επίπεδο. Ήθελα να υπογραμμίσω δύο πράγματα. Το έχω ήδη πει. Όταν δημιουργούμε πλούτο στο τοπικό επίπεδο, απαραίτητα δημιουργείται ένα μικρό προστατευτισμό. Δεν λέω να πάμε κατά των νόμων τη αγορά, αλλά όταν βάζουμε την ανάπτυξη τη υπαίθρου και βάζουμε ε, τα τοπικά χρήματα σε ανταγωνισμό με τα ευρωπαϊκά χρήματα δεν δημιουργούνται ε, συνδέσεις. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ε, με το κοτόπουλο, με τα, όλα τα προϊόντα, με τα εσπεριδοειδή. Πρέπει λοιπόν να δημιουργηθεί αυτός ο πλούτος ώστε οι τοπικές δυνάμεις να μπορέσουν να βρουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν πλούτο όταν δεν υπάρχει τίποτα. Δεύτερο χρειάζεται μια εταιρική σχέση. Σήμερα το πρωί ήδη εγώ επειδή πρόκειται να αποσυρθώ από την πολιτική, δημιούργησα τώρα ένα ταμείο επενδυτικό στην πιο φτωχή χώρα της Αφρικής, στην Κεντροαφρικανική Ένωση. Και η πρώτη δυσκολία που αντιμετωπίζουν είναι οι επιχειρήσεις. Ενώ με τις επιχειρήσεις αυτές έχω εδώ και χρόνια σχέσεις εμπιστοσύνης, μου λένε δεν υπάρχει ασφάλεια. Η εταιρική σχέση λοιπόν είναι αδύνατο να δημιουργηθεί ενώ είναι έτοιμοι ε, να επενδύσουν ε, στην ασφάλεια. Με τις επιχειρήσεις μαζί πρέπει να το κάνουμε αυτό γιατί χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ε, πλούτο γιατί αυτές δίνουν την τεχνογνωσία, υλοποιούν την προσφορά αλλά και τη ζήτηση. Προσφορά και ζήτηση είναι ο παραγόντα κλειδί. Δεν έχει νόημα να δημιουργούμε προσφορά με νέου γεωργού, να του δίνουμε νέε δυνατότητε, αν δεν υπάρχει δομημένη ζήτηση. Ζήτηση καταρχά σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε διεθνέ. Α δούμε την αλυσίδα παραγωγή κρέατος σε κάποιες περιοχές ε, είναι κάποιοι έτοιμοι να αγοράσουν κρέας αλλά για να προαχθεί αυτό το κρέας ε, χρειαζόμαστε μια επιχείρηση και αν η επιχείρηση αυτή δεν λειτουργεί μας λέει δεν έχουμε ασφάλεια ε, πέφτουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Αν λοιπόν διασφαλίσουμε τις συνθήκες ασφαλείας, παρέχουμε εγγυήσεις για την επικινδυνότητα, ίσως να μην είναι το πιο σημαντικό, αλλά θα διευκολύνει σίγουρα τις εγκαταστάσεις κάποιων επιχειρήσεων σε τέτοια μέρη. Το άλλο φυσικά ε, είναι η ολιστική προσέγγιση όπως υπογραμμίστηκε. Πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα στην ολότητα, τους χρειάζεται ε, κατάρτιση, πρέπει να υποστηρίζουμε τις μικρές επιχείρησεις στη Γεωργία, στη Γεωργία, στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία δεν υπάρχει πια τίποτα. Ένα τεράστιο ποσοστό του πληθυσμού πεινάει. Ε, πρέπει λοιπόν να αναδομήσουμε όλη την αλυσίδα παραγωγής, αλλά για να γίνει αυτό Πρέπει να εκπαιδεύσουμε ανθρώπους, να τους καταρτήσουμε, να δημιουργήσουμε τοπικούς συνεταιρισμούς, αλλά να κάνουμε να κινηθεί και η αγορά, οι τοπικές αγορές που πλέον δεν υπάρχουν να τις μετασχηματίσουμε, να τις ηλεκτροδοτήσουμε, να φτιάξουμε δρόμους. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε στην ολότητά τους. Διαφορετικά δεν θα υπάρξει ανάπτυξη. Εγώ ως αρμόδιος ε, της τοπικής ανάπτυξης μιας περιφέρειας έτσι μπορώ να σας πω ότι εργαζόμαστε για την τοπική ανάπτυξη σε τοπικό επίπεδο. Όλα αυτά λοιπόν απαιτούν μια δομημένη προσέγγιση. Η αγορά δεν πρόκειται να τα καταφέρει μόνη της, το υπογραμμίζω. Η μόνη της αγορά δεν καταφέρνει τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν σε τοπικό επίπεδο να ε, εγκαθιδρυθούν κάποιο είδου ταμεία τοπικής ανάπτυξης που συνεργάζονται με τις τοπικές αρχές, τις επιχειρήσεις και το σύνολο των οργανισμών που μπορούν να ε, συμπράξουν για την ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Αλλιώς δεν δημιουργείται πλούτος και όταν δεν δημιουργείται πλούτος έχουμε ένα απίθμενο πηγάδι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τέλος ο κύριος Αρνουλίτσο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσίαση. Άκουσα με πολύ ενδιαφέρον όλα αυτά που είπε ο κύριο Λάντα για την εμπειρία του στον επιχειρηματικό κόσμο όταν μιλάει για τη γεωργία και τη στήριξη. Είναι πολύ ενδιαφέρον το πώς χρησιμοποιούνται τα στοιχεία αλλά και το πώς ε, η γεωργία, ουσιαστικά ποιες επιχειρήσεις ε, ε, θα δραστηριοποιηθούν, τι σπόροι θα χρησιμοποιηθούν, τη διαφοροποίηση, ε, κατά πόσο υπάρχουν διάφορα επίπεδα, ε, πόσες επιχειρήσεις, όταν έχουμε και το πρόβλημα της αρπαγής γης, κατά πόσο υπάρχουν διαφοροποιημένα επιχειρηματικά εγχειρήματα. Θέλουμε ολιστικές ε, λύσεις ε, για την επίτευξη των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, όπως υπόθηκε και από άλλους. Θα πρέπει να πάμε στα Ηνωμένα Έθνη, πιστεύω, και να δούμε πώς χρησιμοποιούνται οι στόχοι βιώσιμης ανάπτυξης. Εσείς είπατε ένα σωρό ωραίους στόχους, εκπαίδευση, διακυβέρνηση, νερό, γεωργία. Ε, ΚΟΠ είπατε στη Βόνη εκεί θα εξετάζουν την γεωργία και το κλίμα και την αλληλεπίδρασή τους εγώ λοιπόν υποστηρίζω να χρησιμοποιήσουμε τους SDG ε, και να δείξουμε σε παρουσίαση όπως τη δική σας τι στόχους έχουμε υιοθετήσει, γιατί θεωρούμε ότι είναι αλληλένδετοι, γιατί πρέπει να προωθήσουμε μαζί με την Κομισιόν στις υπεύθυνη χάραξη πολιτικής ότι τους επιδιώκουμε για κάποιο λόγο. Αύριο θα έχουμε τη συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια όπου θα προσπαθήσουμε να δείξουμε πώς χρησιμοποιούμε τους στόχους βέσμης ανάπτυξης στις πολιτικές μας και για ποιο λόγο. Οπότε αυτή είναι η ερώτησή μου. Μπορούν να, αν είναι να τους εντάξουμε σε μελλοντικέ παρουσιάσεις ποιοι συγκεκριμένοι στόχοι θεωρούνται ε, σημαντικότεροι και πώς ε, ε, συνδέονται μεταξύ τους. Ευχαριστώ και μια γρήγορη ερώτηση από μένα επειδή οι άνθρωποι που θα ζητήσουν αυτή τη χρηματοδότηση να συμμετέχουν σε αυτή τη χρηματοδότηση θα είναι υπάρξουσες επενδυτικές τράπεζες. Αναρωτήθηκα, λοιπόν, Έχουμε κάποια στρατηγική εικόνα του τι είδους επενδύσεις θέλουμε να ενθαρρύνουμε, γιατί ναι, ένα πράγμα είναι οι επιχειρήσεις που θέλουμε να εξάγουν, αλλά απ' την άλλη θα πρέπει να υπάρξει και εσωτερικό, χώρο εμπόριο. Όπως είπατε και εσείς Ρομπέρτο, μιλάμε για εκατομμύρια καταναλωτών που αυτή τη στιγμή δημιουργούνται στην Αφρική και έχουν τις δικές τους εγχώριες αγορές. Νομίζω η αγορά κινητών τηλεφώνων είναι εγχώρια αγορά. Πώς μπορούμε λοιπόν να διασφαλίσουμε... Ήρθε από την Δυτική Όχθη την περασμένη εβδομάδα και εκεί ένα από τα αιτήματα ήταν τέτοιου είδους επενδυτική τράπεζα ε, ιδέες, ε, τι είδους χρηματοδοτήσεις θα γίνουν, να ξέρουν πώς κάνουν οι άλλοι άνθρωποι τα πράγματα ώστε να μην αναφερόμαστε απλά σε εξαγωγές προς εμάς, αλλά στο να δημιουργούνται πραγματικές, αυθεντικές, τοπικές επιχειρήσεις. Ρόμπερτ, έχετε να απαντήσετε σε πολλές ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις έξυπνες ερωτήσεις σας. Όσο εσείς ρωτούσατε, εμείς ε, σημειώναμε τις βελτιώσεις που πρέπει να κάνουμε πριν από τις επόμενες παρουσίες, όχι μόνο για τις αλληλοσυνδέσεις μεταξύ ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης, αλλά και επί της ουσίας. Ας τα πάρουμε με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα το ζήτημα των ε, στόχων βιώσιμης ανάπτυξης. Ε, ε, δεν είναι μόνο τρία τα παραθυρά αυτά, είναι 14-15 νομίζω. Και έχουμε και ένα πίνακα ε, αλληλοσυνδέσεων. Δεν το έχετε δει διότι δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, αλλά πολύ σύντομα θα είναι διαθέσιμο. Παρουσιάστηκε στο Operational Board πριν από δύο-τρεις εβδομάδε. Το πρότυπο μέσω του οποίου όχι οι επενδυτικές τράπεζες αλλά οι αναπτυξιακές τράπεζες θα μας προτείνουν τα προϊόντα τα οποία θα επιλεγούν και περιλαμβάνει στόχους βιώσιμης ανάπτυξης, αριθμό δημιουργίας θέσεων εργασίας, βιωσιμότητα, ποιότητα των θέσεων εργασίας, περιβαλλοντική βιωσιμότητα και όλα αυτά. Όλα αυτά που έχετε συμπεριλάβει στον κανονισμό πολύ σωστά. Όλα αυτά υπάρχουν στο πρότυπο το οποίο θα κυκλοφορήσει αρχές Δεκεμβρίου διότι θα αποτελέσει αυτό το πρότυπο τη βάση πάνω στην οποία οι τράπεζε θα προτείνουν όλα αυτά που θέλουν να κάνουν. Περιλαμβάνει τα πάντα. Είναι αρκετά περίπλοκο, αλλά έτσι χρειάστηκε να γίνουν τα πράγματα. Οι τρει ε, αυτέ φάσει ε, πιστεύω μπορούν να έχουν την υποστήριξή μα. Ε, στην πραγματικότητα, κάθε διαφορετικό προϊόν θα δημιουργηθεί με διαφορετικό τρόπο και θα οργανωθεί διαφορετικά. Αλλά η συμπερίληψη της διατήρησης της βιωσιμότητας είναι κάτι που σημειώνουμε και σίγουρα θα το λάβουμε υπόψη στο πρότυπό μας. Αυτό που είναι σημαντικό είναι τι τους ρωτάει κανείς να του πούν. Δηλαδή μου λέτε θέλετε αυτά τα χρήματα για την εγγύηση, διότι θέλετε να κάνετε 20 χωριά 500.000 ανθρώπων και να βοηθήσετε να δημιουργηθεί η οικονομική ανάπτυξη και η χειραφέτηση εκεί, για παράδειγμα. Η ερώτηση του κυρίου Νόισερ, ε, η δήλωση που μας έκανε, είναι πολύ πρόσδεκτη και λαμβάνω υπόψη το σημείο για την αρπαγή γης που αναφέρατε, που ανέφεραν και άλλοι. Η αρπαγή γης, ε, το land grabbing, Εγώ εξετάζω τους κανόνες, τους εθελοντικούς κανόνες ε, διακυβέρνησης του ΦΑΟ ε, για την ε, κατοχή γης ως συνιστώσεις το μελετάμε. Εγώ θέλω το έγγραφο αυτό να γίνει υποχρεωτικό για τους επενδυτές και για τα προγράμματα που θα εντάσσονται στο επενδυτικό σχέδιο. Δηλαδή προσπαθούμε να εντάξουμε την έννοια της χρηστής διακυβέρνησης όσον αφορά την ιδιοκτησία γης, την έγκαιρη ιδιοκτησία σε σχέση με τις επενδύσεις αυτές, ε, λαμβάνοντας αυτό το έγγραφο που συζητήθηκε και που αποτέλεσε το αντικείμενο διαπραγμάτευσης και να το καταστήσουμε υποχρεωτικό στο πλαίσιο της δέουσας επιμέλειας που θα πρέπει να ε, συμπεριληφθεί σε όλο αυτό. Έχετε δίκιο, το EFSD θα πρέπει να κάνει τη διαφορά ε, για να επιλέγει τους καλύτερους επενδυτές. Ωστόσο πρέπει να σας πω ότι πρέπει να είμαστε καλυμμένοι για τις απώλειες. Αλλιώς, αν πάμε κατευθείαν στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία που αναφέρατε ως παράδειγμα, υπάρχει κίνδυνος να χάσουμε αμέσω όλες τις εγγύσεις. Δεν λέω ότι θα συμβεί σίγουρα, αλλά ο υπολογιζόμενος κίνδυνος βάσει των γνώσεων που έχουμε σήμερα είναι αρκετά υψηλός. Οπότε, αν θέλουμε να μειώσουμε στο ελάχιστο τις απώλειες που θα έχουμε σε δύσκολες χώρες, θα πρέπει να έχουμε κάποια επένδυση σε μια χώρα όπου ο κίνδυνος να χάσει κανείς χρήματα είναι πολύ μικρότερος. Ώστε να μπορούμε να αντισταθμίσουμε με το ποσό που χρεώνουμε για τις εγγύσεις, ε, για παράδειγμα στην Κένια, σε σχέση με αυτό που κάνουμε στο Νότιο Σουδάν. Και ξέρετε, όπως γνωρίζετε, οι σχέσεις αυτές είναι πολύ δύσκολες, όπως είπατε και εσείς κύριε Σαφόζερ. Τώρα για τους συνεταιρισμού. Σίγουρα υποστηρίζουμε και θα το συμπεριλάβουμε ως σύσταση το να υποστηρίζουμε τους συνεταιρισμού. Ωστόσο, όταν μιλάμε για νέα συμμαχία για την επιστημιστική ασφάλεια, εδώ μιλάμε για πολύ ευαίσθητε καταστάσει όπου οι ιδιωτικέ επενδύσει είναι τρομακτικά δύσκολε. Εμεί λειτουργούμε μέσω επιχορηγήσεων, μέσω ΜΚΟ, μέσω ενό ε, συγκεκριμένου δικτύου. Είναι κάτι που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε η μη εμπορική κατάσταση, αλλά αυτή τη στιγμή η ευαισθησία τη κατάσταση είναι πολύ ψηλή. Οπότε η απάντησή μου στο ερώτημά σα είναι ότι σίγουρα ναι, θέλουμε να δημιουργήσουμε ε, ασφαλείς ε, και εξωπρεπείς θέσεις εργασίας και προσπαθούμε να αποφύγουμε, να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της αρπαγής γης ε, στο πλαίσιο των επενδύσεων και φυσικά και μέσω των τοπικών μας αντιπροσωπιών και γραφείων. Τώρα για το μηχανισμό υποβολής παραπώνων το εξετάζουμε. Το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι ε, ουσιαστικά να τρέχει το σύστημα αυτό από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Όποιο αποφασίσει πούμε, να δώσει χρήματα στη Λίντα, αυτή θα πρέπει να είναι το πρώτο σημείο υποδοχή οποιοδήποτε ε, μηχανισμού ε, παραπώνων για την φορολόγηση και τη διαφθορά μπορώ να σας διαβεβαιώσω κατά 100%. Μέχρι στιγμή ε, οι υπηρεσίε τη ταξούντε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή μα έχουν βοηθήσει να αποφύγουμε οποιονδήποτε τέτοιο κίνδυνο και να αποφύγουμε όχι μόνο τι ε, επικίνδυνε ε, δικαιοδοσίες ε, αλλά και τις επικίνδυνες ε, εταιρείε σε ασφαλείς δικαιοδοσίες. Να σας δώσω το παράδειγμα του ε, Μαυρικίου. Όποιος θέλει να κάνει ένα equity fund το πάει να το φτιάξει στο Μαυρίκιο. Εκεί μπορεί να το κάνει κανείς με τρόπο απολύτως αποδεκτό προς εμάς με συγκεκριμένη φορολόγηση, κάποια συγκεκριμένη διαφάνεια και Μπορεί να το φτιάξει όμως με τρόπο που δεν είναι δεκτός ε, ε, για εμάς. Ε, δεν είναι λοιπόν η χώρα το πρόβλημα, αλλά ο τρόπος σύστασης των ιδιών κεφαλαίων του Equity Fund. Οπότε ευχαριστούμε τους συναδέλφους της DigiTaxud που μας βοήθησαν. Τώρα, για διάφορα άλλα πράγματα που ανέφερε ο κύριος Σαφόζερ. Το πρώτο, ο, μικρός, ο μικρής κλίμακας προστατευτισμός. Συμφωνώ. Πράγματι προσπαθούμε όλο και περισσότερο όσο είναι δυνατόν να επενδύσουμε στις τοπικές αγορές υπέρ των τοπικών περιφερειακών αγορών. Η Αφρικανική κοινότητα έχει μια αγορά 160 εκατομμυρίων ανθρώπων με ένα αρκετά εκλεπτισμένο